Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις σας. Θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίσω εγκάρτια στην συνάντηση αυτή. Έχουμε μια καλή συνήθεια εδώ, σύμφωνα με την οποία τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό οργανώνουν τέτοιες συναντήσεις για σημαντικά θέματα και μάλιστα που έχουν μακροπρόθεσμα μεγάλη σημασία Σήμερα και αύριο λοιπόν θα συζητήσουμε την περίπτωση της εφαρμογής ενός New Deal για την οικονομική αναθέρμανση την ανάκαμψη της Ευρώπης. Με μεγάλη χαρά λοιπόν καλωσορίζω τον πρόεδρο Σομπότκα της Γερουσίας της Τσεχίας που κάθεται αριστερά μου, δεξιά μου μάλλον. Καλωσορίσατε κύριε πρόεδρε και επίσης με μεγάλη χαρά Βλέπω εδώ και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Τσεχίας, τον κύριο Βούλτσεκ. Αριστερά μου έχω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον Επίτροπο Αλμούνια, τον οποίο επίσης καλωσορίζω Συχνά δεχόμαστε επιτρόπους και χαιρόμαστε κάθε φορά ιδιαίτερα που ο πρόεδρος της Κομισιόν αυτή τη φορά και επίση και ο Επίτροπος Αλμούνια έρχεται πολύ συχνά μαζί μας. Επίσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα θα έρθει περίπου στις 5 και 20 Υπήρξαν πολλά προβλήματα στην ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρώπη σήμερα και καθυστερήσεις. Στις 3.25 συγγνώμη θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα, επομένως θα ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Jean-Claude Trichet, ο οποίος δεν είναι ακόμα παρόν. Ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι σύντομα μαζί μας. Θα σας πρότεινα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του κυρίου Αλμούνια και στη συνέχεια συνέχεια θέλετε να πείτε εσείς κάτι προηγουμένως. Εσείς θα ξεκινήσετε πρώτα. Αναφέρετε στον κύριο Σομπότκα, κύριο Πέτρη. Vážené dámy, vážení přátelé, kolegyně, kolegové, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα στην εισαγωγή μου να δηλώσω καταρχάς ότι ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης είναι μια φυσική αντίδραση που βασίζεται ακριβώς στην αντίληψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη οικονομικά σταθερή, ανταγωνιστική ως προς τον υπόλοιπο κόσμο, μια Ευρώπη που να μην ελέγχεται από μια χούφτα προνομιούχων γραφειοκρατών αλλά που να είναι φιλική προς όλους τους πολίτες της. Και με βάση τις αρχές αυτές θέλουμε να αντιδράσουμε. Η ελεύθερη κυκλοφορία βέβαια των ανθρώπων, των εμπορευμάτων και του κεφαλαίου είναι κάτι που δεν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε. Σήμερα που αντιμετωπίζουμε μία σφαιρική κρίση πρέπει οι ειδικοί οικονομολόγοι αλλά και εμείς οι πολιτικοί να αντιδράσουμε και να συμμετάσχουμε στο καθήκον της αντιμετώπισης της με βάση την αρχή που σας ανέφερα. Απλούστερα δηλαδή, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να γίνει με τους ίδιους λογικούς κανόνες που ακολουθούσαμε και πριν ξεσπάσει η κρίση. Βέβαια πρέπει να πάρουμε ορισμένα μαθήματα για να αποφύγουμε στο μέλλον τα λάθη που οδήγησαν σε αυτήν την κρίση. Αλλά δεν πρέπει να υποκύψουμε στον πανικό. Γιατί η λύση, η αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι ο προστατευτισμός και η ναπολεόντια στάση ορισμένων ηθινόντων. Η, μια Ευρωπαϊκή Ένωση με δύο ταχύτητες με βάση τη διατήρηση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των παλαιών και νέων χωρών μελών δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε αρνητικές εμπειρίες όπως η σχεδιασμένη οικονομία του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ. Όταν, αν χάσουμε την πίστη μας στις αρχές μας, θα καταλήξουμε σε πειραματισμούς και τυχοδιοκτισμούς και δεν θα βρούμε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν η Ευρώπη μπορεί να παίξει έναν ουσιαστικό και στρατηγικό ρόλο. Αν αντί να δημιουργεί χιλιάδες γραφειοκρατικές οδηγίες δεν πρέπει μάλλον να επικεντρώσει την προσοχή της στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που να λειτουργεί με βάση την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της γεωργίας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το μέλλον αν λάβουμε τα μέτρα αυτά. Η Ευρώπη διαθέτει αρκετούς οικονομολόγους ώστε να μπορέσει να βρει μια τη λύση στην κρίση. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και πολλοί λαοπλάνοι και γραφειοκράτες που θα θελήσουν να υποφεληθούν από την κρίση για να εξυπηρετήσουν τους εγωιστικούς τους στόχους. Αν καταφέρουμε όμως να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να πετύχουν στα κακόβουλα σχέδιά τους. Δεν πρέπει βέβαια να ζητήσουμε, να αποκλείσουμε την κριτική. Δεν θέλουμε να φημώσουμε όσους διαφωνούν. Απλώς εγώ παραμένω αισιόδοξο ότι η Ευρώπη θα καταφέρει με κοινή προσπάθεια όλων των κρατών να διατηρήσει τη θέση της στον κόσμο και μάλιστα και να την ενδυναμώσει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. So much, uh, President Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σομπότκα και τώρα έχει το ρόλο ο κύριος Βούλτσεκ. Κύριε Πρόεδρε Πέτεριν, κύριε Πρόεδρε Σομπότκα, αγαπητοί Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, χαίρομαι, τιμή είναι για μένα που είμαι εδώ σε αυτή την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση. Δεν είναι για μένα αυτό μία δραστηριότητα μάλιστα ανιεροί συνηθισμένη στα πλαίσια ε, της Προεδρίας μας σε προηγούμενους μήνες συμμετείχα σε συναντήσεις με συναδέλφους και εξέτασα σημαντικά θέματα και θέματα επίλυσης των προβλημάτων ύφεση. Εδώ λοιπόν ανάλογα με τον προσανατολισμό των διαφόρων ομάδων και να δούμε και τα επίκαιρα θέματα. Η οικονομική δημοσιονομική κρίση η παγκόσμια κατέληξε να γίνει μια βαθιά ύφεση οικονομική και μετά και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουμε την επανεμφάνιση αυτής. Δυστυχώς διαδίδεται, εξαπλώνεται και από την ε, άσχημη ρύθμιση της αμερικανικής ε, οικονομίας. Βλέπουμε μια μείωση της ζήτησης προϊόντων, ε, μια πολιτική που δεν είναι η σωστή όπως πρέπει. Βλέπουμε διάφορες απειλές που εμφανίζονται για μια ηθική επίσης κρίση και αυτό επηρεάζει την σκέψη μας, τους λογισμούς μας αυτή η φέση οικονομική και με τις δυνάμεις αγοράς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή και επίσης να δούμε πώς μέσω των φόρων θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε την κατάσταση από κοινωνικής πλευράς. Βλέπουμε μια τρομερή κρίση βέβαια και εθνικισμούς οικονομικούς. Βλέπουμε και ναζιστικό κίνδυνο, φασιστικό κίνδυνο λόγω της ύφεσης αυτής. Ο κόσμος, οι πολίτες χάνουν πια την πίστη ακόμα και στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζονται ενέργειες από πλευράς Οικονομικής Ένωσης ε, και εμείς καταδικάζουμε τις λύσεις που περιορίζονται στα σύνορα των εθνικών κρατών. Χρειάζεται ένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε από κοντά τα αίτια της κρίσης. Μια κοινή πολιτική για μια ανάκαμψη, αναδιοργάνωση της αγοράς και αποτελεσματικά μέτρα. Επίσης μια συντονισμένη πολιτική απέναντι σε όσους δεν επιθυμούν να κάνουν τίποτα, να λάβουν τίποτα σαν μέτρα και απλά και μόνο υποφεληθούν από τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη-μέλη. Βέβαια, θα πρέπει να ίσως να δούμε και πώς θα πληρωθούν αυτά τα λάθη στα πλαίσια μιας ρύθμισης. Χρειάζεται μια σταθεροποίηση των ε, ε, αγορών αλλά δεν είναι μόνο ότι πρέπει να πληρώσουμε τα σπασμένα. Χρειάζεται μια αποκατάσταση εμπιστοσύνη ε, στα ε, στους φορείς ε, και νομίσαμε ότι το πρόβλημα θα το έλυνε η αυτορύθμιση αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται μια ρύθμιση με απαιτητικά μέτρα. Είναι όλα αυτά ρυθμίσεις που δεν είναι τέλειες βέβαια αλλά είναι απαραίτητες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει καλύτερα την ποιότητα αυτών των ρυθμίσεων στο μέτρο στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης και ότι χρειάζεται μια ολοκλήρωση αυτών των μέτρων στα πλαίσια των κρατών μελών και στις ΗΠΑ ε, τα προβλήματα αυτά επιτάχυναν την παγκόσμια κρίση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερες ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε ε, να επηρεαστεί κατάλληλα η κατάσταση, όχι περισσότερη ρυθμίση, περισσότερα μέτρα, αλλά αποτελεσματικότερα μέτρα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη ζήτηση. Επίσης, θα ήθελα να χαιρετήσω τα πρώτα βήματα που έγιναν προς την σωστή κατεύθυνση και ένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισμός αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί τίθεται και ένα θέμα σήμερα το ερώτημα μήπως έφτασε η ώρα να έχουμε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και να υποστηρίξουμε οικονομικά. Ε, σημειώνουμε μια καθυστέρηση στις επενδύσεις, στις νέες τεχνολογίες ε, και πολλοί είναι που εγκαταλείπουν το σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σχολεία πολύ νωρίς είτε αποφυτούν να από κακά σχολεία. Θα πρέπει να προλάβουμε μια μελλοντική κρίση, λύνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα της σημερινής κρίσης. Επίσης, περισσότερο για την ασφάλειά μας χρειάζεται η κατάλληλη υποδομή δική μας ε, και να καλύπτονται οι ενέργειες μας. Θα πρέπει να δούμε νέους στόχους που θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Η ευρωπαϊκή μας οικογένεια θα πρέπει να προσπαθήσει να πετύχει μια συνοχή για να ξεφύγει από τη δαγκάνη αυτής της κρίσης. Και ίσως η κρίση είναι και μια δοκιμή για την υπομονή μας, για τις ικανότητές μας να ξεφύγουμε, για να προωθήσουμε νέες ιδέες και καινοτομίες τεχνικές. Ε, το κάθε κράτος αν μείνει απομονωμένο θα είναι αδύναμο για να επιλύσει παρόμοιες κρίσεις ενώ το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι κάτι το ισχυρό που θα μπορούσε να λύσει αυτά τα προβλήματα. 27 κράτη μαζί είναι το πιο, ο πιο ισχυρός συνασπισμός στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να λύσουμε τα προβλήματα που προκαλούν την κρίση. Και όλα αυτά θα πρέπει να συγκλίνουν σαν μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή μας σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε Βέλτσεκ. Από τα σχόλια και των δύο παρεμβενόντων βλέπουμε ότι υπάρχουν σημεία έμφαση τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα να πω από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι έχουμε εμπιστοσύνη μεν καταρχήν στην αγορά αλλά λέμε ότι η αγορά χρειάζεται και μια κάποια ρύθμιση και η συνθήκη της Λισαβόνας έχει σαν κέντρο της την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δηλαδή ότι η αγορά δεν είναι αυτός σκοπός. Η αγορά πάντα πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και θα πρέπει επομένως να βασιζόμαστε στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για να εκφράσουμε αυτή την αντιμετώπιση. Εγώ τώρα θέλω να καλέσω να δώσω το λόγο σε κάποιον ο οποίος ήταν παρόν στην συνάντηση των 7 βιομηχανικών χωρών στη Ρώμη, πάντα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι παρόν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζουακίν Αλμούνια για να παρουσιαστεί και στο απόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε Πέτερινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ευρωκοινοβούλιο. Προσκάλεσε την Κομισιόν και εμένα προσωπικά να πάρω σε αυτή εδώ τη συζήτηση. Εκ μέρου τη Κομισιόν, λοιπόν, καλωσορίζω και εγώ του εθνικού βουλευτέ και του προέδρου των ε, Άνω και Κάτω βουλής στο Τσεχικό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με αυτά που είπανε. Η Ευρώπη έχει μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αντιμετωπίζουμε μια μοναδική οικονομική κρίση. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε αυτή την κρίση, να τη φανταστούμε πριν από 1,5 χρόνο όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, ότι σήμερα δηλαδή θα αντιμετωπίζουμε μια βαθιά ύφεση στις οικονομίες μας. Την Παρασκευή, αμέσως πριν ξεκινήσει η συνάντηση των G7 στη Ρώμη, η Eurostat έδωσε τα νούμερα για το ΑΕΠ των χωρών μας. Τέλος 2008. Δυστυχώς τα νούμερα αυτά ήταν στο μείον. Λίγο χειρότερα από τα νούμερα που προβλεπόντουσαν προβλέψαμε εμείς τις προβλέψεις μας στις 19 Ιανουαρίου μείον 1,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 2008. Αναγωγή. Και αυτό δείχνει ότι μπαίνουμε φέτος σε ύφεση στην Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2009 και η Αμερικάνικη οικονομία μπαίνει σε ύφεση. Το ίδιο και η Ιαπωνία. Τα νούμερα στην Ιαπωνία για το τέταρτο τρίμηνο του 2008 τα είχαμε και είναι ακόμα χειρότερα από τα αμερικάνικα και τα ευρωπαϊκά νούμερα. Πριν από μερικούς μήνες ακόμα συζητούσαμε αν ήταν δυνατόν να γίνει αποσύζευξη. Δηλαδή συζητούσαμε ακόμα πριν από μερικούς μήνες μόλις τη δυνατότητα για αναδυόμενες οικονομίες να μπορέσουν να κρατήσουν μια ανάπτυξη αρκετά ισχυρή και να λειτουργήσουν ως ατμομηχανή στην παγκόσμια οικονομία έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την ύφεση. Δυστυχώς όμως η κινέζικη οικονομία, η βραζιλιάνικη οικονομία, η οικονομία της Ινδίας βέβαια ακόμη έχουν μια κάποια ανάπτυξη ωστόσο και αυτές υποφέρουν από επιβράδυνση και όλες οι αναδυόμενες οικονομίες και αυτές έχουν αρνητική ανάπτυξη. Και το παγκόσμιο εμπόριο που δείχνει την αλληλεξάρτησή του ανάμεσα στις βιομηχανοποιημένες οικονομίες από τη μια, τις αναδυόμενες οικονομίες από την άλλη, των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών και των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών, οι δεσμοί μειώθηκε το παγκόσμιο εμπόριο με μεγάλη ταχύτητα από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα. Μάλλον μέσα στο 2008 μέχρι σήμερα. Καθολική λοιπόν η κρίση. Άρα, τι βλέπουμε, η παγκοσμιοποίηση μας έδωσε πολλές ευκαιρίες, ωφεληθήκαμε από το μεγάλο, μεγαλύτερο βαθμό αλληλεξάρτησης των οικονομιών μας, την τελευταία φάση του κύκλου. Τώρα όμως έχουμε τον αρνητικό αντίκτυπο στην κρίση των βιομηχανικών χωρών προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και όλοι αρχίζουν να υποφέρουν από κοινωνικές εντάσεις, κοινωνικές συγκρούσεις ως συνέπεια της ε, οικονομικής επιβράδυνσης. Ποια ήταν η ευρωπαϊκή μας αντίδραση. Ως Ένωση είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια αυτή κρίση. Με την έννοια ότι συντονίζουμε τις οικονομικές πολιτικές μας, έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό. Έχουμε την Κεντρική Τράπεζα και ο κύριος Τρισέ σε μερικά λεπτά θα είναι εδώ. Μπορεί να μιλήσει αυτός για τις αποφάσεις και το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά και άλλες κεντρικές τράπεζες και στην Ευρώπη και έξω από τα σύνορα της Ένωσης αντέδρασαν συντονισμένα όσον αφορά ε, την, νομισματική πολιτική. Έτσι ώστε να υπάρξει ρευστότητα για το σύστημα πιο πολύ από ό,τι γινόταν σε παρελθούσες καθολικές υφέσεις έτσι ώστε νομισματικά ήμασταν σε θέση να αντιδράσουμε. Όσον αφορά τη δημοσιονομική μας πολιτική, επίσης έχουμε μάθει στην Ευρώπη να συντονίζουμε τις δημοσιονομικές μας πολιτικές. Η συνθήκη από το Μάστριχτ και μετά ορίζει ένα ε, πλαίσιο συντονισμού και προσανατολισμού των δημοσιονομικών πολιτικών παρότι οι δημοσιονομικές πολιτικές παραμένουν κυρίως ε, της αρμοδιότητας των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων ωστόσο υπάρχουν κανόνες για δημοσιονομική πειθαρχία το δημοσιονομικό πλαίσιο η σύγκληση, το σύμφωνο σταθερότητας η συζήτηση όλων αυτών των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ, η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, όλα αυτά ήταν χρήσιμα, χρήσιμα εργαλεία και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ύφεστα εργαλεία αυτά για να συντονίσουμε τη δημοσιονομική μας αντίδραση και ως συνέπεια αυτού του συντονισμού η Κομισιόν πρότεινε και το το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε πέρυσι προς το τέλος του χρόνου το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης European Recovery Plan. Η δημοσιονομική πολιτική που να χρησιμοποιείται με αντικυκλικό τρόπο, με διακριτικό τρόπο και έτσι οι Ευρωπαίοι απάντησαν συντονισμένα. Αυτό είναι θετικό, πολύ θετικό. Το ότι οι πρωθυπουργοί όλων των χωρών μας κατάφεραν να συμφωνήσουν για μια κοινή αντίδραση. Και τώρα αρχίζουμε να αξιολογούμε, να κάνουμε έναν απολογισμό. Ποια ήταν η επίπτωση αυτής της αντίδρασης στις οικονομίες μας. Αρχικές εκτιμήσεις. Και τις επεξεργαζόμαστε όλο και περισσότερο. Θα τις παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το, το Μάρτιο. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις μας, η διακριτική αυτή η δημοσιονομική τόνωση που αποφασίστηκε από τα κράτη-μέλη της Ένωσης τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι ισοδύναμη περίπου με το 1% του ΑΕΠ. Επίσης πάρθηκαν και εθνικές αποφάσεις για επιπλέον ε, δημοσιονομικά κίνητρα στην οικονομία 0,5% επιπλέον και στην Ευρώπη σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι αυτόματοι σταθεροποιητές. Εκτιμούμε ότι η επίπτωση αυτών των αυτόματων σταθεροποιητών προκειμένου να τονωθεί η οικονομία ισοδυναμη μεταξυ μεταξύ 2009-2010 περίπου το 1,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Συνολικά λοιπόν, ως άθροισμα, η υποστήριξή μας δημοσιονομικά με αυτόματους σταθεροποιητές και με την διακριτική παρέμβαση είναι ανάμεσα στο 3,3 με 4% του ΑΕΠ φέτος και του χρόνου. Τρίτη ομάδα μέτρων κατά της κρίσης. Η υποστήριξη στις τράπεζες, στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μέτρα προκειμένου να λειτουργεί ομαλά, να, οι χρηματαγορές να λειτουργούν και όλα τα ιδρύματα εκεί που, που, πάσχουν άμεσα από την κρίση σε συντονισμό πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κοινέ κατευθυντήριες γραμμές εγγυήσεις που δόθηκαν και από εθνικές κυβερνήσεις προς τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα στην κάθε χώρα. Έχουμε κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για την επανακεφαλοποίηση, κεφαλαιοποίηση των ιδρυμάτων αυτών και με ιδιωτικό χρήμα και με δημόσιο χρήμα και στις δύο περιπτώσεις οι κοινέ κατευθυντήριες αυτές γραμμές στοχεύουν στο να κρατηθούν δίκαιοι κανόνες του παιχνιδιού για όλους. Αποφάσεις που μπορούν να παρθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική μας αγορά. Δεν μπορούν να αποτελούν άνηση μεταχείριση ανάμεσα σε ένα α χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και σε ένα β. Ούτε να υπάρξει άνηση μεταχείριση μεταξύ μιας χώρας μέλους και μιας άλλης χώρας μέλους. Παρακολουθούμε και εποπτεύουμε την εφαρμογή των διαφόρων αυτών υποστηρικτικών πακέτων προς το χρηματοπιστωτικό τομέα μέσα στα πλαίσια αυτά των κατευθυντήριων γραμμών και αρχίζουμε να συζητούμε, όπως ξέρετε, ε, τι να γίνει με στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι επισφαλή διότι ακόμα και με τα μέτρα αυτά όλα τα μέτρα που ανάφερα η πιστοληπτικές αγορές δεν λειτουργούν ομαλά. Πρέπει να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της ρευστότητα της πίστης όσο πιο σύντομα γίνεται και στην Ευρώπη και στις Πολιτείες και σε άλλες οικονομίες αν δεν αποκατασταθεί μια ομαλή κατάσταση στην αγορά πιστώσεων ούτε η νομισματική πολιτική μπορεί να σταθεί ούτε το δημοσιονομικό πακέτο και η υποστήριξη θα είναι αποδοτικό. Αυτό είναι το τρίτο λοιπόν βήμα το συζητάμε. Το Σεββατοκύρικο στην ε, G7 στη Ρώμη το συζητήσαμε και με τους Ιαπωνέζους και με τους Αμερικάνους πώς είναι δυνατό να συντονίσουμε τη δράση μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα-πρώτα όμως πρέπει να αποφασίσουμε μεταξύ μας. Αυτό θα είναι το κλειδί για τις επόμενες εβδομάδες. Και στην άτυπη συνάντηση των Πρωθυπουργών την 1η Μαρτίου αυτό θα συζητηθεί. Αυτό είναι με πρωτοβουλία της Ιχικής Προεδρίας όπως ξέρετε πώς θα προετοιμαστεί η ευρωπαϊκή θέση έναντι της επόμενης συνάντησης των G20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου. Οι φορολογούμενοι έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και κοιτάνε. Λένε ναι, κατανοούμε ότι οι τράπεζες, ο τραπεζικός τομέας πρέπει να λειτουργεί. Κατανοούμε ότι η πιο μεγάλη πρόκληση, η επίγουσα πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τις χρηματοπιστωτικές αρχές είναι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των χρηματογορών. Χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να βγούμε και να μπορέσουμε να βγούμε από την ύφαση. Αλλά αυτά τα λεφτά του φορολογούμενου που παίρνουν σε κίνδυνο με την υποστήριξη αυτή προς το χρηματοπιστωτικό κλάδο απαιτεί διαφάνεια. Έχουν το δικαίωμα να ξέρουν, να ξέρουμε τι υπάρχει πίσω από τον ισολογισμό κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Απαιτούνται σκληροί όροι για τους μάνατζερς, τους διευθυντές που, πρέπει να που θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της τράπεζας και που ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό και στο παρελθόν. Απαιτούνται συστήματα να αποφευθεί η αντικυκλική δράση ή μάλλον η κυκλική δράση σε σχέση και με τις ανάγκες σε κεφάλαιο και όσον αφορά τις αμοιβέ των ε, ανωτάτων στελεχών, χρηματομεσητών επίσης, και διαφάνεια. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό θέμα, ένας πολιτικός όρος που θα συνοδεύει την μεταφορά πόρων προς το χρηματοπιστωτικό τομέα τις εβδομάδες που έρχονται θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα παρακολουθούμε να δούμε ποια είναι η πραγματική επίπτωση του των δημοσιονομικών πακέτων στην οικονομία μας. Στο πρόγραμμα ανάκαμψης η σύστασή μας είναι να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για το πακέτο αυτό, να γίνεται εγκαίρος και να γίνεται στο σωστό χρόνο. Τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν αν θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι καλό στην προσπάθεια αυτή όσον αφορά την δημόσια παρέμβαση με λεφτά του φορολογούμενου. Ταυτόχρονα, παράλληλα δηλαδή με την παρακολούθηση του πώς εφαρμόζεται αυτό, πώς υλοποιούνται αυτά τα κίνητρα, παρατηρούμε ότι σε μερικές χώρες υπό την εποπτεία και της Κομισιόν και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οικονομίες μερικών κρατών μελών τις παρακολουθούν ιδιαίτερα στενά οι αγορές. Μερικά spread στα κυβερνητικά ομόλογα αυξάθηκαν πολύ τους τελευταίους μήνες ή τον τελευταίο 1,5 μήνα και αυτά τα spread, αυτές οι διαφορές των επιτοκίων, η αύξηση της διαφοράς του spread δείχνει, αποκαλύπτει ότι σε σχέση με τον δημόσιο οικονομικά μεταξύ των κρατών μελών η θέση δεν είναι η ίδια. Αυτό μας θυμίζει ότι η βιωσιμότητα είναι ύψης της σημασίας για όλους και αυτό μας θυμίζει ταυτόχρονα ότι ναι μεν δίνουμε ένα δημοσιονομικό, μια τόνωση, ένα κίνητρο για να έχουν περισσότερη ζήτηση που μόνο ο δημόσιο τομέα με τη δημοσιονομική του πολιτική μπορεί να δώσει στι σημερινέ συνθήκε, ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά, να υπαγρυπνούμε, μην βάλουμε σε κίνδυνο την μέσο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Και γι' αυτό η εφαρμογή του δημοσιονομικού μας πλαισίου, του Συμφώνου Σταθερότητας, είναι ιδιαίτερα σημαντική στις σημερινές συνθήκες. Με το σύμφωνο αυτό, μετά την αναθεώρηση του 2005, η αναθεώρηση αυτή του 2005 έδωσε περισσότερη ευελιξία δράσης στα δημόσια οικονομικά στις κακές στιγμές του οικονομικού κύκλου. Τη χρειαζόμαστε αυτή την ευελιξία τώρα. Ταυτόχρονα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να συνδυάσουμε αυτή την ευελιξία με μια αυστηρή απέτηση μέσω μακροπρόθεσμης σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών για να μην βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον των οικονομιών μας και να μην βάλουμε σε κίνδυνο ε, τις επόμενες γενιές. Η Ευρώπη θα μας βοηθήσει να βγούμε σιγά σιγά από την καταιγίδα αυτή. Η Ευρώπη είναι ένα καταφύγιο. Παρέχει προστασία η Ευρώπη. Σε μερικά άρθρα Διαβάζεται οι λεγόμενοι αναλυτές, οι εμπειρογνώμονες εντός εισαγωγικών συζητάνε το ενδεχόμενο η Ευρωζώνη να διασπαστεί. Η πιθανότητα γι' αυτό είναι μηδέν. Σας το λέω, μηδέν. Σαφώς μηδέν. Αλλά οι υποψήφοι για να μπουν στην Ευρωζώνη τους επόμενους μήνες και χρόνια, ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Πιο μεγάλος είναι ο κατάλογος αυτών που θέλουν να μπουν από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Το ευρώ είναι ένα εργαλείο προστασίας μας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτές τις κρίσεις. Αλλά το ευρώ επίσης απαιτεί ευθύνη για όλα τα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και αυτή η ευθύνη κυρίως αναφέρεται στο πώς κάθε χώρα μέλος αντιμετωπίζει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μέσω μακροπρόθεσμα. Και μία τελευταία λέξη, όπως είπα και πριν, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ευρωπαϊκή συζήτηση και οι ευρωπαϊκές λύσεις της Ένωσης ενώ Θέλουμε να δώσουμε και μια ευρωπαϊκή συμβολή στην παγκόσμια λύση που θα βρεθεί στη συνάντηση 2 Απριλίου στο Λονδίνο των G20 ή στις συζητήσεις που τα διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα ε, οργανώνουν την Άνοιξη μετά το Λονδίνο. Έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση της Διεθνούς Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει. Η Ευρώπη συμβάλλει στην αναζήτηση καθολικών λύσεων, παγκόσμιων λύσεων και η Ευρώπη πρέπει να το κάνει με μία φωνή, με μία θέση, με σαφείς ιδέες. Έχουμε συμβάλει αρκετά από την αρχή της διαδικασίας αυτής των παγκόσμιων ε, ε, συνεδριάσεων στην Ουάσινγκτον και αλλού θα το κάνουμε και στο Λονδίνο και ελπίζω τα δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια, το άτυπο 1η Μαρτίου και το επίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 19 Μαρτίου και πιο πριν η συνάντηση των Ευρωπαϊκών Μιλών του G20 και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα την επόμενη Κυριακή στο Βερολίνο, όλα αυτά θα δώσουν σαφή μηνύματα πώς μπορούμε να συμβάλλουμε να βρεθεί μια παγκόσμια λύση. Ένα στοιχείο συμβολής, μια παράμετρος και επενώ ιδιαίτερα την Τσεχική Προεδρία για την σαφή θέση που παίρνει. Μία συμβολή λοιπόν, μία από τις πιο σημαντικές θα έλεγα, εκ μέρους της Ένωσης για την παγκόσμια λύση των κρίσεων είναι η ανάγκη να αποφύγουμε τον προστατευτισμό. Να προστατεύσουμε την εσωτερική μας αγορά, να προστατεύσουμε τους πολίτες μας έναντι του κινδύνου προστατευτισμού και να συμβάλλουμε στο να υπάρξει μια παγκόσμια οικονομία ανοιχτή με ελεύθερη κυκλοφορία εργασίας, προσώπων, προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων. Και είναι αλήθεια ότι αυτές οι ελευθερίες που είναι ουσιώδεις πρέπει να συναδεύονται από υπαρκή ρύθμιση. Αλλά αυτός ο συνδυασμός μεταξύ ελευθεριών και ρύθμισης θεωρώ ότι δεν υπήρχε όταν δημιουργήθηκαν οι σημερινές ανισορμέρειες, ανισορροπίες. Και θα πρέπει να αποτελέσει στοιχείο για να βρεθεί λύση για τις κρίσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Θα πρότεινα τώρα, επειδή ο πρόεδρος Τρισέ δεν έχει καταφτάσει ακόμα, να ζητήσω από τους δύο εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρουσιάσουν την έκθεσή τους και θα το διακόψουμε ή όταν τελειώσετε θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον πρόεδρο Τρισέ παρουσιάσει την απόψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά από τους δύο εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουμε δύο εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δύο προς ένα για να έχουμε μια ισορροπημένη συζήτηση. Θα δώσω λόγο λοιπόν στον Κλάους ε, Λένε και μετά την κυρία Έρτσοκ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, θα ήθελα να σας τονίσω ότι αυτή η συνάντηση έχει μια πολύ σημαντική λειτουργία σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει από το 2005 μια ομάδα διευθυντική κατά κάποιο τρόπο, μια ομάδα κατεύθυνσης που προετοιμάζει τις διασκέψεις κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αυτό είναι και μια μορφή συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία της Λισαβόνας. Εγώ χαίρομαι για το γεγονό ότι σήμερα βλέπω τόσου πολλού εθνικού κοινοβουλευτικού στην αίθουσα αυτή για να μπορέσουμε να ανταλλάξουν απόψει μαζί μα και να παρουσιάσουν τη δική του άποψη για την προετοιμασία τη Εαρνή Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φυσικά το κυρίαρχο θέμα είναι η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι αντίθετα με την προηγούμενη πρακτική του στο παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένα θέματα όπω παραδείγματο χάρη ενεργειακή πολιτική, αλλά κυρίω στο ζήτημα του πώ θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την οικονομική κρίση. Και εδώ, όταν μιλάμε για ένα New Deal στην Ευρώπη, αυτό έχει πολλού λόγου να χρησιμοποιούμε αυτή την ε, διατύπωση, γιατί αυτή η κρίση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο σημασία και έκτασης που μπορεί να συγκριθεί μονάχα με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τέλος της δεκαετίας του 20 και την αρχή δεκαετίας του 1930 και ήταν γνωστά ως η Μεγάλη ύφεση. Και ο πρόεδρος Ρούσβελ των ΗΠΑ είχε την ιδέα του λεγόμενου New Deal, <clears throat> της νέας μοιρασιά, της νέας αντιμετώπισης, να προχωρήσει με μια πραγματιστική ιδεολογία, να προχωρήσει για να αντιμετωπίσει την ε, ανάγκη επίλυση μια σοβαρή οικονομική κρίση. Πρέπει να σα πω λοιπόν ότι και σήμερα η κατάσταση δεν είναι διαφορετική από την κατάσταση τη δεκαετία του 1930 και γι' αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε κι εμεί με ένα είδο New Deal για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα ενώπιό μα. Αυτό όμω σημαίνει ότι πρέπει να πούμε εκπεφρασμένα ότι δεν θα πρέπει να γυρίσουμε, να επαναχωρήσουμε στην εποχή πριν από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Δεν θέλουμε προστατευτισμό, δεν θέλουμε υπερχρέωση, θέλουμε να διατηρηθεί το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Φυσικά με του μηχανισμού ευκαμψία που προσφέρει, θέλουμε να έχουμε μια πραγματιστική στοχοθεσία για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτή την κρίση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και του εθνικού ε, των εθνικών συστημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα χρήματα που έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο συντονιστού. Δεν θα πρέπει μια κρίση η οποία αντιμετωπίζεται σε ένα κράτος με ένα αλφα τρόπο να οδηγήσει σε κρίση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία και εγκαλείται να προσφέρει λύσεις. Να εξασφαλίσει ότι στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει μια συμβολή στο να αποφύγουμε την επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης στο μέλλον, να μειώσουμε την πιθανότητα επανάληψης και θα σταθούμε και στο θέμα αυτό. Εγώ θέλω να κάνω τώρα εξής μια συγκεκριμένη παρατήρηση. Νομίζω <clears throat> ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες στον κόσμο σε σχέση με άλλες οικονομίες και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια και μέσω της διαδικασίας της Λισαβόνας έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Γι' αυτό η Ευρώπη και η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναζητήσει στη διαδικασία της Λισαβόνας την συνέχιση των απαντήσεων για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της ε, ε παγκοσμιοποίησης. Και αυτό πρέπει να πούμε σαφώς εν ώψη της ε, συνόδου ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση γιατί έχουμε κάνει σημαντικές συμβολές για το θέμα αυτό. Έχουμε επίσης και τη θεματική του ευρώ. Όλοι και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε και στο ψήφισμα, θα πρέπει να χαιρόμαστε για το γεγονό ότι υπάρχει το ευρώ. Γιατί το ευρώ έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουμε να έχουμε συνθήκε στην Ευρώπη οι οποίε είναι σχετικά θετικέ παρά την κρίση στον κόσμο. Και έχουν παραμείνει σταθερέ και σχετικά θετικέ οι συνθήκε στην Ευρώπη. Φανταστείτε πώ θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε ακόμα τα εθνικά νομίσματα αν έπρεπε κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση σε μια χώρα να ξεσπάσει μια τραπεζική κρίση με όλα τα προβλήματα αστάθειας τα οποία προκύπτουν από κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κατανοήσουμε και να λεχθεί σαφώς το ψήφισμά μας ότι χάρη στην επιλογή του ευρώ έχουμε επιτύχει να βελτιώσουμε πάρα πολύ την κατάσταση. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε συνάδελφε. Επειδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κύριος Τρισέ δεν έχει προσέλθει ακόμη θα δώσω το λόγο στην κυρία Έντιθ Χέρτσοκ Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Σοσιαλιστικής Ομάδας και θα ήθελα να τονίσω το ανθρώπινο πρόσωπο που έχει και πρέπει να έχει κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ανακλέγεται άμεσα από τους πολίτες είναι το καταλληλότερο όργανο για να την αντιμετωπίσει. Καθώς ξέσπασε η συνολική σφαιρική χρηματοπιστωτική κρίση φάνηκε ότι η Ευρώπη και οι πολίτες της πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει το δρόμο παγκόσμια. Να αυξηθεί η απασχόληση και να παταχθεί η μαζική ανεργία. Να αποφύγουμε τον προστατευτισμό που συνοδεύει συνήθως και τον εθνικισμό. Και για να αποφευθεί να αντιμετωπιστεί η κρίση λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε την κοινωνία της γνώσης και να δώσουμε στους πολίτες την ασφάλεια που χρειάζονται. Πρέπει να συνδέσουμε τα χρηματοπιστωτικά κίνητρα που μπορούμε να δώσουμε με άλλους τομείς που τονίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας, όπως την ενέργεια, την έρευνα, την καινοτομία. Τα εργαλεία που χρειάζεται η Ένωση για να εφαρμόσει τους στόχους της Λισαβόνας είναι βασικά η απλοποίηση όλων των προγραμμάτων. Όλα τα εργαλεία και νομοθετήματα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να ξεσπάσει νέα κρίση. Βέβαια αν εφαρμοστούν διαφορετικά και πολλά εθνικά σχέδια θα είναι βέβαιο, το μόνο βέβαιο είναι, θα είναι ότι θα ξεσπάσει και νέα κρίση πρέπει αντίθετα η Ένωση να δράσει ως ένα σώμα. Οι μακροοικονομικές ανισότητες δεν είναι μόνο κάτι το χρηματοοικονομικό αλλά κρίση του συστήματος στο υποφίλεται σε κοινωνικές ανισότητες μεταξύ άλλων και στην έλλειψη κανονισμών και κανόνων. Μόλις άρχισε να φαίνουν, άρχισαν να φαίνονται οι αρνητικές συνέπειες της έλλειψης αυτής κανόνων και διακανονισμού. Θα κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Όπως και το 89 έχω το αίσθημα ότι η κατάσταση αλλάζει μέρα με τη μέρα και εμείς δεν, δεν την αντιμετωπίζουμε. Οι σοσιαλιστές λοιπόν πιστεύουν ότι ο μόνος δρόμος για να ξεφύγουμε από την κρίση είναι να λάβουμε μέτρα από και για τους λαούς. Να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες απασχόλησης και να αποφευθεί η μαζική ανεργία. Αυτός ο στόχος πρέπει να καθορίζει να είναι το ύψιστο κριτήριο για το λεγόμενο νέο New Deal για την Ευρώπη. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρηματοδοτήσει προγράμματα κυρίως επαγγελματικής μετεκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το κύριο θέμα είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Βέβαια, αφορά και τους εργοδότες, ιδίως των μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως είπε και ο Δαρβίνος πριν από 200 χρόνια, η θεωρία της φυσικής επιλογής δεν σημαίνει ότι το δυνατότερο ή το ισχυρότερο είδος θα επιβιώσει, αλλά το πιο έξυπνο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να δώσουμε την πιο έξυπνη δυνατή απάντηση στην πρόκληση αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει αυτόν τον δρόμο να επιλέξουμε, αυτή να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, να είμαστε εμείς οι εξυπνότεροι. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί ένα σύστημα να φανεί εξυπνό, μόνο οι άνθρωποι μπορούν. Πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν τον έλεγχο των τραπεζικών συστημάτων ή έναν πιο θεσμοθετημένο καπιταλισμό να υπάρξει ως δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία αλλά ταυτόχρονα και ασφάλεια για τους πολίτες. Πρέπει να υπάρξει καινοτομία ώστε οι οικονομίες μας να γίνουν πιο παραγωγικές και να συνδέσουν τους πολίτες με το πολιτικό σύστημα. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ανοίξουν περισσότερο τις αγορές των τηλεπικοινωνιών και το βιομηχανικό τομέα ιδιαίτερα η Ευρώπη Μπορεί λοιπόν να βγει από αυτήν την οικονομική διαταραχή και να αποτελέσει, να παίξει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της. Σημαντικό εκτός από την αύξηση της παραγωγικότητας είναι και η παιδεία. Πρέπει η παιδεία και η διαβίου μάθηση να αποτελέσουν προτεραιότητες. Γιατί έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα με την δημιουργία των καταλήλων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους. Συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θέλουν να τονίσουν το θέμα των πολιτών και του λαού, διότι μόνο μέσω και για τον λαό μπορεί η Ευρώπη να ευημερήσει. Αυτή είναι, αυτό είναι το σοσιαλιστικό μας όραμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τα λόγια σας. Και τώρα καλώς ήρθατε στον διοικητή της ε, Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, τον Ζακλό Να σε ενημερώσω ότι όσοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο στην όλη συζήτηση θα πρέπει να το ζητήσουν προηγουμένως. Θα έχουμε πάντα δύο ομιλητές, επαναλαμβάνουμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο καθένας θα έχει δικαίωμα για τρία λεπτά. Το λόγο έχει ο, Ζαν Κλωτρισέ. Κύριε Πρόεδρε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Γερουσίας και του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας Τσεχίας, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εδώ συμμετέχω στις Βρυξέλλες σε αυτή τη συνάντηση. Μέσα Φεβρουαρίου μόνο, αλλά είναι η τρίτη μου συνάντηση φέτος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια τώρα αυτή τη φορά. Τρίτη φορά λοιπόν, τι δείχνει ότι ο διάλογος ανάμεσα στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Κοινοβούλιο είναι πραγματικός και στενός. Σας γυρίσω στα γερμανικά. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας εξαιρετικής κατάστασης. Η παγκόσμια οικονομία νιώθει μια σημαντική συγκυριακή κάμψη. Αυτό έχει συμπεριλάβει, αυτό το γεγονός έχει συμπεριλάβει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες έχουν αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση με αποφασιστικότητα και θέλω να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο για μένα φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Ότι μέσα στην ενωμένη μας αντιμετώπιση δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να τον ίσο ενώπιον σας. Ένας από τους πρώτους μας στόχους λοιπόν ως πολιτικοί λήπτες αποφάσεων είναι να επιλύσουμε αυτή την κρίση σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίε οι οποίες βρίσκονται πίσω από αυτή την κρίση, τις αιτίε του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, στις μακροοικονομικές πολιτικές των κυριωτέρων παικτών και στην διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική. Πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι οι σημερινές μας αποφάσεις δεν προετοιμάσουν ανάλογε επαναλήψεις του φαινόμενου αυτού στο μέλλον. Και επομένω η κύρια μου πρόταση σήμερα είναι ότι αν μπορέσουμε να χαράξουμε πολιτικές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επανέλθουμε στο status quo ante, αλλά αντίθετα ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία έχει τη σωστή εστίαση για να εξασφαλίσουμε μέσω πρόθεσμα τη σταθερότητα, τότε μπορούμε να αποτρέψουμε κρίση στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό. Η παγκόσμια οικονομία ήταν και εξακολουθεί να είναι και σήμερα χωρίς ισορροπία σε τρεις τομείς. Στο χρηματοοικονομικό σύστημα, στις μακροοικονομικές συλλήψεις και αντιμετωπίσεις των κυβερνήσεων και στην διακυβέρνηση τη χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονική τη παγκόσμια οικονομία. Η κρίση αυτή δεν μα δίνει μονάχα μια δυνατότητα επανεξισορρόπηση, μα δίνει την υποχρέωση να επανεξισορροπήσουμε του τρει αυτού αλληλένδετους τομεί τη παγκόσμια οικονομία. Δεν πρέπει να αποτύχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού τους τρεις τομείς όσο και δύσκολο να είναι το έργο το οποίο θα χρειαστεί για την αντιμετώπιση του να σας τονίσω που νομίζω ότι είναι πιο έντονες αυτές οι προκλήσεις ξεκινώντας από τις αιτίε της κρίσης. Είναι σαφές ότι η αιτία της κρίσης ήταν η μαζική υποεκτίμηση των κινδύνων σε, στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα όλων των μεγάλων οικονομιών. Λόγω της χρηματοοικονομικής καινοτομία φτάσαμε να έχουμε αδιαφανείς διαδικασίες στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη αύξηση του βιωτικού επίπεδου, σε μια μείωση των ε, ε, spreads, των διαφορών μεταξύ των αποδόσεων των ε, αξιογράφων και επίσης σε μια παρότρινση για μαζική αγορά ακινήτων και άλλων στοιχείων του ενεργητικού. Όλα αυτά με την λαθασμένη εντύπωση ότι θα εξακολουθούν να αυξάνονται στο διηνεκέ οι τιμέ των στοιχείων των ενεργητικού και των ακίνητων και ότι δεν υπήρχαν πια οικονομικοί κύκλοι. Αλλά η κρίση μας έδειξε πόσο μη ρεαλιστικοί ήταν αυτές οι ιδέες. Η οικονομική οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι είχαν μεγάλο μοχλοβραχίωνα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έπεσαν θύμα αυτής της κρίσης. Επίσης οι μακροοικονομικές πολιτικές έχουν διαδραματίσει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε πολλές οικονομίες γιατί δεν ήταν αρκετά εστιασμένες στη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα και στην αηφορία των οικονομιών γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει μακροοικονομικές ελλείψεις ισορροπίας οι οποίες ισορρεύτηκαν. Και όλα αυτά πάλι οφείλονται στη λαθασμένη εντύπωση ότι σε μια παγκοσμιωμένη οικονομία, μερικές χώρες θα μπορούσαν με βέλτιστο τρόπο να δανείζονται από άλλες χώρες ή να δανείζουν άλλες χώρες σε έναν τρόπο ο οποίος θα συνέχιζε στο διενεκές. Αυτό μπορεί να οδήγησε σε μια ταχεία οικονομική μεγέθυνση, αλλά τελικά αποδείχθηκε μια λαθασμένη αντιμετώπιση, γιατί η κρίση τελικά οδηγεί του επενδύτε να φοβούνται του κινδύνου και αυτό εμποδίζει και τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει, αλλά και ολόκληρε οικονομίε να αποστρέφονται την χρέωση και την καινοτομία. Έχουμε λοιπόν επίσης και πολλά προβλήματα διακυβέρνησης της οικονομίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν πολλά ψεγάδια ακόμα στη διεθνή οικονομική αρχιτεκτονική. Δεν είναι εδώ το πρόβλημα μιας λανθασμένης ή υπεραισιόδοξης εκτίμησης. Απλώς φάνηκαν τα προβλήματα στη διεθνή συνεργασία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συντώνησε μία παγκόσμια διαβούλευση για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες της παγκοσμίας αγοράς στους G7. Οι G7 έχουν τονίσει επίσης επανειλημμένα τα προβλήματα ελλείψεως ισορροπίας. Υπήρξαν πολιτικές προτάσεις και κατευθύνσεις οι οποίες έχουν προταθεί και εγκριθεί αλλά δεν εφαρμόστηκαν πλήρως σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης δεν φάνηκε ο κίνδυνος διαφθοράς και διάβρωσης του πλαισίου αυτό. Θέλω να τονίσω ότι οι κεντρικές τράπεζες ήταν αυτές οι οποίες έκαναν τις πιο σαφείς δημόσιες δηλώσεις για την ανάγκη ο δημόσιος τομέας να προετοιμαστεί για σημαντικές διορθώσεις στην πορεία του σε ό,τι αφορά την αγορά. Αυτό ήταν το μήνυμα της ε, συνάντησης της Βασιλείας το 2006 των κεντρικών τραπεζών και επίσης στην αρχή του 2007. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία μέσω της δικής της έρευνας ήταν αυτή η οποία υπήρξε η πιο διαυγής σε σχέση με τα προβλήματα αυτά από όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα με ποιο τρόπο θα ανακτήσουμε την ισορροπία στο διεθνέ χρηματοοικονομικό σύστημα, στι μακροοικονομικές πολιτικέ και στην διακυβέρνηση του οικονομικού τομέα. Για το χρηματοοικονομικό σύστημα χρειάζονται πιο αυστηρέ ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσει θα πρέπει να αποτρέψουν μια επανάληψη των υπερβολών που είδαμε στι χρηματαγορές και θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα και μια προοπτική σταθερότητα. Το Φόρουμ σταθερότητα έχει ήδη εντοπίσει του κύριου χώρους όπου χρειάζεται να υπάρξει μεταρρύθμιση, τρεις δυο τομείς όπου είναι απαραίτητη η αλλαγή κατά την άποψή μου. Πρώτον, το να εισάγουμε κίνητρα και κανόνες για να μην εστιάζεται υπερβολικά ο χρηματοοικονομικό τομέα στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο και μόνο. Δεύτερον, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το επίπεδο των κινδύνων στο χρηματοοικονομικό σύστημα και σε ό,τι αφορά του ε, φορεί, τι αγορέ και τα εργαλεία που είναι ή χωρίς ρύθμιση ή ανεπαρκώς ρυθμισμένα και τρίτον να εξαλείψουμε όπου αυτό είναι εφικτό τα στοιχεία τα οποία μεγενθύνουν την τάση του χρηματοοικονομικού συστήματος να σωρεύει υπερβολικά υψηλό κίνδυνο και να μην λειτουργεί σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή να μειώσουμε το θετικό feedback της κυκλικής λειτουργίας οικονομίας. Όλα αυτά αναφέρθηκαν και στο ανακοινωθέν των G7 που δημοσιεύτηκε το, Σάββατο, το περασμένο Σάββατο και δεν πρόκειται να τα αναφέρω όλα αυτά, αλλά σήμερα θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γενικό πλαίσιο της μακροοικονομικής πολιτικής για το μέλλον. Γιατί είναι απαραίτητο, γιατί είναι επιτακτικό, βραχυπρόθεσμα να υπάρξει σταθεροποίηση της τωρινής κατάστασης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε από τους οφθαλμούς μας την ανάγκη να έχουμε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική η οποία θα σταθεροποίηση τις οικονομικές συνθήκες και θα αποτελεί βάση για τις μελλοντικές προσδοκίες τόσο σε εθνικό όσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δούμε λοιπόν την κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα, υπάρχουν μέτρα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά τα οποία εφαρμόστηκαν με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή και Κεντρική Τράπεζα ήταν μια από τους πρώτους φορείς οι οποίοι αντέδρασαν με την παρακολούθηση της χρηματαγοράς όταν φάνηκαν για πρώτη φορά τα δείγματα μιας επερχόμενης κρίσης το καλοκαίρι του 2007 σε ό,τι αφορά την πολιτική επιτήρησης η κατευθυντήρια γραμμή μας ήταν πάντα να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των δημόσιων στην περιοχή του ευρώ στο μεσοπρόθεσμο επίπεδο βάσει του ότι η αύξηση της ε, νομισματικής μάζας θα πρέπει να είναι, ο πληθωρισμός μάλλον θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο 2%. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν στοχεύαμε να εξασφαλίσουμε τη συνολική σταθερότητα της περιοχής του ευρώ. Αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητο να μην μας οδηγήσουν οι πολιτικές μας στις ανισορροπίες που είδαμε στο παρελθόν, διότι αυτές οι ανισορροπίες ήταν αυτές οι οποίες προξένησαν και οδήγησαν στην σημερινή κρίση. Δεν πρέπει οι λήπτες αποφάσεων να εστιάζονται μονάχα σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, θα πρέπει αντίθετα να αντιμετωπίσουν το πιο μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα με το στόχο του να εξασφαλίσουμε μια σταθερή και μόνιμη ανάκαμψη. Οι σωστέ λοιπόν πολιτικέ δράσει περιλαμβάνουν δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το να έχουμε μια αξιόπιστη στρατηγική εξόδου που θα είναι αντικείμενο σχεδιασμού και σωστή εφαρμογή από τη στιγμή που τα μακροοικονομικά μέτρα έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα και δεύτερον, οι πολιτικές δεν πρέπει να έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση μονάχα, αλλά να δημιουργήσουν και τις απαραίτητες μακροχρόνιες διαρθρωτικές αλλαγές. Περιτώ να σας πω ότι τα στοιχεία αυτά ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ισχύουν και για την Ευρώπη. Οι πολιτικές υπέρ της σταθερότητος είναι απαραίτητος για να αντιμετωπιστεί η κρίση και η κρίση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη να ακολουθήσει η Ευρώπη αυτή την οδό της σταθερότητα. Εμεί θα πρέπει να χαιρόμαστε για το γεγονό ότι η Ευρώπη στο παρελθόν έχει ακολουθήσει μια τέτοια σόφρονα στατιστική και να μην την απολέσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική, οι διεθνεί φορεί θα πρέπει να πείσουν τι χώρε να αναλάβουν πολιτικέ οι οποίε κατευθύνονται προ τη σταθερότητα και να εξασφαλίσει ότι λαμβάνουν υπόψη τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα όπου τα αυτά είναι απαραίτητα και οι διεθνεί χρηματοοικονομικοί φορεί επίση θα πρέπει να, να προσαρμόσουν τη δράση του. Αυτό σημαίνει ότι όπως οι κεντρικές τράπεζες έχουν τροποποιήσει τη στάση τους με διεθνή συνεργασία, με παγκόσμια συνεργασία των κεντρικών τραπεζών που αντανακλά την παγκοσμιοποίηση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να το πράξουν το ίδιο και τα παγκόσμια χρηματοδοτικά όργανα. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας με μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα στο μέλλον από ό,τι τώρα την ε, σχέση μεταξύ μακροοικονομικής σταθερότητας και πολυμερούς επιτήρησης. Μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ φορέων όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το άτυπο όργανο που είναι το Διεθνές Φόρουμ Σταθερότητας θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρειάζεται να βελτιώσει την επιτήρησή της και την χρηματοοικονομική επιτήρηση σε ό,τι αφορά τα, τις χώρες οι οποίες έχουν συστημική σημασία στο παγκόσμιο σύστημα. Εμείς έχουμε τονίσει την ανάγκη επιτήρησης αναδειωμένων και αναπτυσσομένων οικονομιών, αλλά οι βιομηχανικές χώρες θεωρούν ότι είναι άμμο μέσα από τέτοιου είδους επιτήρηση και παροχή συμβουλών. Αλλά η κρίση μας έδωσε πραγματικά ένα μάθημα ότι και οι βιομηχανοποιημένες οικονομίες χρειάζονται και αυτές επιτήρηση των οικονομιών τους, μια αυστηρή επιτήρηση των οικονομιών τους. Όλοι οι παγκόσμιοι φορείς, όλα τα παγκόσμια φόρα θα πρέπει να σκεφτούν για το πώς θα μπορέσει να βελτιωθεί αυτή η επιτήρηση και η αποτελεσματικότητά της για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές πολιτικές. Είναι ένα μακρό μακρό, ένας μακρός και δύσκολο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και δεν έχουμε ακόμα άλλε απαντήσει αλλά η Ευρώπη μπορεί να δραματίσει ένα σημαντικό και ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε πολιτικές που στοχεύουν στη σταθερότητα με μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση μέσα στην Ευρώπη και μπορούμε έτσι να προωθήσουμε καλύτερη διεθνή συνεργασία για να μπορέσουν αυτέ τι πολιτικέ να ακολουθηθούν και από άλλε χώρε σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένω έτσι να αποτρέψουμε μια επαναφορά του status quo ante και πάλι σα λέω ότι η κρίση αυτή μα δίνει την υποχρέωση να τροποποιήσουμε τι βασικέ αιτίε των ανισορροπιών στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα αλλά και σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία της μακροοικονομικής πολιτικής στις χώρες μας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε διοικητά της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση όπως σας είχαμε πει ο κύριος Ζασίντου από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ομιλητές και να τους συγχαρώ. Αναφέρουν όλες οι παρεμβάσεις τις κοινέ ανησυχίες μας σε σχέση με το εγχείρημα που μας εμπλέκει όλους, τις πολλαπλές διαστάσεις αυτής της κρίσης που θα πρέπει να μάθουμε να τις αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να μάθουμε να βρίσκουμε τις λύσεις για όλα αυτά. Έχουμε μια χρηματοοικονομική κρίση, μια οικονομική κρίση, μια κοινωνική κρίση, αλλά και μια πολιτική κρίση. Όλα αυτά με ε, ένα περίγραμμα το οποίο είναι ασαφές και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα μας οδηγήσει, αλλά με σαφείς κινδύνους να προκύψουν πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της μέλη, για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ανανέωση στην πολιτική μας και μια στεναρή πολιτική. Να υπάρχει ένα νέο πολιτικό όραμα, μια νέα λογική ότι δεν πρέπει η συνολική αντιμετώπιση των παγκοσμιοποιημένων θα πρέπει να μας οδηγήσει να ξεχάσουμε το τοπικό στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη και μια συνοχή μεταξύ της συνολικής παγκόσμιας αντιμετώπισης και της δράσης σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ισχυρή ηγεσία, ένα ισχυρό συντονισμό σε όλα τα επίπεδα για να αποφευχθούν ταραχές και συγκρούσεις στο κοινωνικό επίπεδο και επίσης για να μπορέσει να ρυθμίσει με έναν τρόπο αποτελεσματικό μια σειρά προβλημάτων τα οποία συνάπτονται με τη μορφή των χρηματοοικονομικών διαστάσεων φορέων μάλλον σε διεθνές επίπεδο και προβλημάτων. Εδώ θα ήθελα να θέσω στον κύριο Επίτροπο, αλλά ο κύριος Επίτροπος δεν είναι πια παρόν. Ίσως κάποιος άλλος από τους παρεμβαίνοντες θα είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ε, συνθήκης της μεταρρυθμιστικής της Λισαβόνας όπως έλεγε το προηγουμένως. Όταν συζητείται αυτή η συνθήκη είχαν λεχθεί πολλά για τη σημασία που είχε αυτή η συνθήκη για να μπορέσει η Ευρώπη να αρθρώσει το λόγο της και να ορθώσει το ανάστημά της ως ένας παίκτη σε διεθνές επίπεδο. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία μας αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και το ερώτημα που θέλω να θέσω στους ομιλητές είναι τι πιστεύετε για την μεταρρυθμιστική συνθήκη της συνθήκης της Λισαβόνας, πώς μπορεί αυτή η συνθήκη να συμβάλλει στην επιλύση, των προβλημάτων αυτών για τα οποία συζητούμε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και θα... κάποιος θα σας απαντήσει σίγουρα. Έντμοντ Βίμπροτ ε, από την Πολωνική Γερουσία. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οργάνωση της συνάντησης αυτής. Για το θέμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει αυτό το σύνθημα η Ευρώπη χωρίς σύνορα, χωρίς εμπόδια μάλλον γιατί εδώ βρισκόμαστε μπροστά μια, σε μια παρόμοια κρίση και μίλησαν ε, και από τη Βουλή και από τη Γερουσία για το θέμα αυτό ε, από την ε, Δημοκρατία της Τσεχίας. Εδώ θέλουν να κλείσουν τις αγορές εργασίας. Εμφανίζονται εθνικισμοί καινούργοι λοιπόν και αναφέρεται και μεταβατική περίοδος μακρύτερη για το άνοιγμα της αγοράς εργασίας. Όπως επίσης ε, για ε, μεταφορά δραστηριοτήτων από άλλες χώρες σε αυτή τη χώρα. Εδώ δεν θα πρέπει κανείς να διπλωθεί στον εαυτό του. Θα πρέπει να ανοιχτεί περισσότερο με περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Βέβαια, κάνοντας το χρέος μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν κράτη-μέλη. Δεύτερο σημείο όλες αυτές οι ανησυχίες που ισχύουν ε, και για την Πολωνία επίσης είναι με ποια μέτρα θα ξεπεράσουμε αυτή, αυτή την κρίση αλλά να μην είναι το φάρμακο χειρότερο ε, από το σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε. Ίσως μπορούμε να βρούμε τη λύση, τη θεραπεία μας χωρίς το φάρμακο αυτό. Δεν για προστατευτισμούς κλπ. Αλλά είμαστε κατά των προστατευτισμών αυτών γιατί θα μπορούσε να υπονομεύσει την οικονομία της αγοράς με διάφορες ε, επιδοτήσεις το ένα το άλλο, βοήθειες ε, σε διάφορους τομείς και όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα σε άλλα κράτη-μέλη και κυρίως αν θέλει κανείς να βοηθήσει, να επιδοτήσει και παλιούς οικονομικούς τομείς τότε τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε με τις, με τις καινούριους τομείς ε, τις καινοτομίες επίσης τι θα γίνει με όλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι είναι κάτι το βασικό να σεβαστούμε το σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας πέρα βέβαια από αυτό που είπε επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από λίγο. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι να εξυπηρετούν τους πολίτες, να μας χαρακτηρίζουν μια ισορροπία στη λήψη μέτρων και επίσης σε σχέση με τα όσα είπε ο Επίτροπος κ. Σαλμόνια. Οι υπεύθυνοι των όσων συνέβησαν θα πρέπει να υποστούν και τις συνέπειες γιατί στην Πολωνία όταν κοιτάζουμε την τηλεόραση ή στις Βρυξέλλες επίσης βλέπουμε πολλές διαφημίσεις ναι προσφέρουμε δάνεια ε, το ένα τ' άλλο εύκολα μάλιστα αλλά τι γίνεται, τι καταλάβαμε από όσα έχουν συμβεί αν έχουμε παρόμοιες διαφημίσεις Ευχαριστώ ναι, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Γκούναρα Έκμαρ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, τις μέρες που ζούμε ακούμε την φράση «χρειάζεται δράση». Διαφωνώ όμως με αυτό. Θα ήθελα να πω τώρα είναι η στιγμή για σωστή δράση. Right action που σημαίνει ότι οι πράξεις μας θα πρέπει να συμφωνούν με τους κανόνες και τα θεμέλια που φέρουν μαζί σε ένα σύνολο της οικονομίας και της χώρας μας. Και αυτό ισχύει και όταν συζητάμε και τις χρηματαγορές ή όταν συζητάμε τις κρατικές ενισχύσεις και την διατήρηση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό. Διότι αν στρεβλώνουμε τις αγορές σε μία χώρα, τις υπονομεύουμε τις αγορές και σε άλλη χώρα. Και το βλέπουμε αυτό στις χρηματαγορές. Και το βλέπουμε αυτό σε κάθε πλευρά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αν δεν τηρούμε τους κανόνες, κάνουμε ζημιά σε άλλους. Και η ηρωνία και το παράδοξο εδώ είναι ότι νομίζουμε ότι ωφελούμαστε, ότι ωφελεί τη δική μας οικονομία, ενώ στην πράξη υπονομεύοντας τις άλλες οικονομίες σε ένα κόσμο που όλοι εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον. Να το πω αλλιώ. Αν στρεβλώσουμε τον ανταγωνισμό και αν έχουμε λιγότερο εμπόριο, αυτό θα σημαίνει και λιγότερες εισαγωγές αλλά και λιγότερες εξαγωγές. Και οι σύγχρονες οικονομίες ζουν ουσιαστικά με αυτό. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση όπου χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Και ένα ισχυρότατο μήνυμα από αυτή την κοινή μας σημερινή κοινοβουλευτική συνάντηση πρέπει να είναι ότι δεν δεχόμαστε προστατευτικά μέτρα. Γιατί κάνουν ζημιά σε όλους μας. Τα προστατευτικά μέτρα σε μία χώρα κάνουν ζημιά σε όλες τις άλλες 26 χώρες. Και τελικά όλοι ανήκουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις 26 χώρες. Οι 26 συν μία. Εξάλλου ο προστατευτισμός συνήθως και πάντα θα έλεγα προηγείται του εθνικισμού και υπονομεύει την ενοποίηση που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Ας είμαστε λοιπόν σαφείς στο μήνυμά μας. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει διέξοδος και λύση με πολιτικές που χρησιμοποιούν κρατικές ενισχύσεις ή καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό και έλεγχο των δημόσιων οικονομικών. Έλλειψη ελέγχου, συγγνώμη, των δημόσιων οικονομικών η Ευρώπη δεν χρειάζεται προστατευτισμό. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και τώρα είναι η στιγμή για σωστή δράση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και τώρα το λέγω έχει ο επόμενος ομιλητής, ο Χρήστος Παπουτσής από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει αιτίες. Αιτίες στις οποίες αναφέρθηκε προηγουμένως τόσο ο κύριος Τρισέ όσο και ο κύριος Αλμούνια. Αιτίες οι οποίες όμως αφορούν ορισμένες από τις βασικές παραδοχές της κυρίαρχης ιδεολογίας. Και αν αυτές τις αιτίες δεν τις, δεν τις αποσαφηνίσουμε, εάν δεν προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αυτές τις αιτίες, φοβάμαι ότι θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και η κρίση θα είναι μπροστά μας στα επόμενα χρόνια. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η επόμενη μέρα της κρίσης θα είναι εντελώς διαφορετική όπως επίσης χρειάζεται να αναζητήσουμε τις λύσεις με διαφορετικά εργαλεία με διαφορετικές μεθόδους. γι' αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πρώτα απ' όλα σε μια νέα αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά όσον αφορά την ευρωπαϊκή ένωση και σε μια νέα αρχιτεκτονική του κοινοτικού προπολογισμού. γιατί όταν μιλούμε για, την δημοσιονομικά, για τα δημοσιονομικά για τη δημοσιονομική θεωρία είναι απολύτως βέβαιο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αντικυκλική πολιτική και αναρωτιέμαι τι είδους αντικυκλική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιήσει η ευρωπαϊκή ένωση χωρίς μια αναθεώρηση των βασικών προτεραιοτήτων και των δομών του κοινοτικού προϋπολογισμού. γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε νέες προτεραιότητες νέες επιλογές πρώτα απ' όλα όσον αφορά το ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων δεύτερον όσον αφορά το μοντέλο της ανάπτυξης που χρειαζόμαστε και τρίτον όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού και των κρατικών προμηθειών. Και σε αυτό επιμένω γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για παράδειγμα στις νέες απαιτήσεις της εποχής μας όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη εάν η επιλογή μας όσον αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών της ένωσης δεν αφορά τις νέες τεχνολογίες που οθούν, που δίνουν μια νέα όθηση στην πράσινη ανάπτυξη, δεν αφορούν την εκπαίδευση των εργατών, των εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να μετεκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες της πράσινης ανάπτυξης και επιπλέον δεν θα δημιουργήσουμε και νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές πρέπει πράγματι να εστιαστούν στη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα και στην αηφορία αλλά πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να πάρουμε και τις απαραίτητες πολιτικές επιλογές σε σχέση με τους στόχους που θέλουμε να έχουν οι πολιτικές μας. Και εγώ σπέβδω να πω ότι χρειαζόμαστε πολιτικές τέτοιες οι οποίες να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, χρειαζόμαστε πολιτικές που να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να ενισχύουν το κοινωνικό κράτος και ταυτόχρονα να φέρνουν στην αγορά στην αγορά τους μηχανισμούς της ρύθμισης και της εποπτείας. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα έδειξε ότι η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών. χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανισμού ρύθμιση και εποπτεία των αγορών όπω επίση και μηχανισμού για, το τραπεζικό σύστημα ούτω ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. γι' αυτό και θα ήθελα να ακούσω τον κύριο τρισέ εάν θα μπορούσε πράγματι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να περιλάβει στη στρατηγική τη το θέμα τη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση ω βασικού στόχου για την επικέντρωση των πολιτικών τη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την Πολωνία. Ναι. Θα ήθελα με τη σειρά μου να πω ότι χρειάζεται να λύσουμε αυτή την κρίση την οικονομική και έχουμε νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια απειλή για την κοινωνία μας, για τις κοινωνίες μας, αλλά είναι και μια ευκαιρία για ένα καινούριο άνοιγμα. Θα πρέπει εμείς οι πολιτικοί να βοηθήσουμε για μία έξοδο από την κρίση αυτή και έτσι να ενισχυθούμε αντί να αποδυναμωθούμε θα πρέπει οι νέες να μην είναι εις βάρος της ενιαίας αγοράς, να μην είναι εις βάρος των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είναι εις βάρος της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης της ίδιας. Πιστεύω επίσης ότι μετά και από όσα εδώ υπόθηκαν ότι χρειάζεται ένας ορίζοντας κοινό. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά οι εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη δρούν εντελώς διαφορετικά, ενεργούν διαφορετικά. Μιλάμε για προστατευτισμό, γιατί είδαμε μέτρα προστατευτικά. Και λυπάμαι που ένας εκπρόσωπος από μια από τις ε, μεγαλύτερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λέει ότι ναι, θα ενισχύσει την εθνική του βιομηχανία εάν κλείσουν οι θηγατρικές των ξένων Τι γίνεται, αυτός είναι αντάξιος της ιδέας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαθέτουμε ένα πραγματικό ηγέτη Ευρωπαίο. Δεν έχουμε μια καινούρια ιδέα, θαραλέα ιδέα στην Ευρώπη. Οι προτάσεις για να ξεφύγουμε από την κρίση αυτή θα πρέπει να έχουν διάσταση ευρωπαϊκή. Χωρίς μια ευρωπαϊκή διάσταση θα καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει τεράστια σημασία. Είναι πολύ σπουδαίο τώρα λίγο πριν και από τις ευρωεκλογές. Οι υποψήφοι στις ευρωεκλογέ θα πρέπει να εξηγήσουν ποιες είναι οι προθέσεις τους, ε, τι θα ήθελαν, πώς θα ήθελαν να βοηθήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να υπερασπιστούν τα όσα έχουμε ήδη πετύχει. Θα πρέπει να μας μιλήσουν για προοπτικές ανάπτυξης και όχι μόνο πώς θα ξεφύγουμε από αυτήν τη σκοτεινή σύραγγα σε επίπεδο εθνικό ή τοπικό. Αυτό ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει Ρόμπερ Γκέμπελ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τρία λεπτά μπορώ να κάνω μόνο μερικά σχόλια. Θα ήθελα να πω πρώτον ότι ζούμε μια κρίση σφαιρική του συστήματος. Είναι γνωστό το φαινόμενο από τους ασχολούμενους με την πληροφορική. Κάθε σύστημα έχει αδύνατα σημεία και αυτά αυξάνονται όσο αυξάνονται οι διασυνδέσεις. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται στο επίπεδο του συστήματος ολόκληρου. Αυτό έγινε και στην παγκοσμιοποιημένη χρηματοπιστωτική διαδικτύωση. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει. Πρώτα να αποφύγουμε τα ψεύτικα προβλήματα και ένα από αυτά είναι η πιθανολογούμενη καταστροφή του συστήματος του ευρώ. Νομίζω ότι ο Επίτροπος Αλμόνια το είπε πολύ καλά, τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Το ευρώ κατά τη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης υπήρξε προστασία όχι μόνο για την Ευρωζώνη αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Αντίθετα, νομίζω ότι πραγματικό πρόβλημα είναι η ένταση που αυξάνεται μέσα στην εσωτερική αγορά μετά από τις λανθάνουσες υποτιμήσεις ορισμένων νομισμάτων σε σύγκριση με το ευρώ όπως την Βρετανική Λύρα που υποτιμήθηκε κατά πάνω από 20%. Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι να καταπολεμήσουμε τη... τον πειρασμό του να στραφεί ο καθένας προς τον εαυτό του δηλαδή να καταπολεμήσουμε τον προστατευτισμό και να ενισχύσουμε το συντονισμό των μακροοικονομικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι τώρα έχει επιτυχώς εφαρμόσει την πολιτική της, μείωσε ορισμένα επιτόκια, αλλά άλλες τράπεζες δεν καταφέρνουν να μεταφέρουν τη μείωση αυτή των επιτοκίων σε όφελος των πελατών τους. Δύο τρίτα μάλιστα των τραπεζών έχουν γίνει πιο απαιτητικές και πιο αυστηρές ως προς τη χορήγηση δανείων. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Κατά δύο τρίτα μειώθηκαν τα δάνεια που τους χορηγούν. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει αναθέρμανση. Φυσικά τα εθνικά σχέδια Καλά είναι, ιδίως εάν χρηματοδοτηθούν χωρίς υψηλά δάνεια. Αλλά η Ευρώπη θα έπρεπε ακόμη περισσότερο μέσω της ε- Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να λάβει μέτρα. Το κεφάλαιο της αυξήθηκε πρόσφατα μέσω της χρησιμοποίησης ορισμένων αποθεμάτων, αν όμως και τα κράτη βάζανε λίγο το χέρι στην τσέπη από τα εθνικά τους προγράμματα για να αυξηθεί το κεφάλαιο της ΕΤΕ θα μπορούσε αυτή να κάνει περισσότερες προσπάθειες υπέρ των επιχειρήσεων και αυτό νομίζω ότι θα ήταν η εκδίκηση του Προέδρου Τρισέ. Δεν θα ήταν επιστροφή στο status quo. Αυτά είχα να σας πω σύντομα συνάδελφοι. Σίγουρα δεν είναι πλήρη, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνάντηση και τη συζήτηση αυτή, διότι η κρίση έδειξε ότι οι στόχοι της Λισαβόνας ήταν σωστοί και ότι τα κράτη που έκαναν τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τους επιτύχουν είναι και εκείνα που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, έλαβαν το λόγο και μάλιστα σεβάστηκαν το χρόνο ομιλίας Τώρα έχουμε προβλέψει την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών ε, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Καλάζεκ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο θα ήθελα εδώ με την ευκαιρία να χαιρετήσω την παρουσία των Προέδρου της Γερουσίας και του Κοινοβουλίου της ε, Δημοκρατίας Τσεχίας, επίσης ε, και τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κύριο Τρισέ. Χαίρομαι που τον βλέπω εδώ μαζί μας ε, και είμαι περήφανος που σήμερα λαμβάνω το λόγο εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα βέβαια να ζητήσω συγγνώμη που θα πρέπει αμέσως μετά να εγκαταλείψω την αίθουσα γιατί θα πρέπει για το 2007 την απαλλαγή από τον προϋπολογισμό να μιλήσω γι' αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συγγνώμη λοιπόν θα αναγκαστώ να αποχωρήσω. Αλλά στα όσα σύντομα θα πω θα ήθελα να πω μερικά πράγματα ακριβώς για την όλη δύσκολη σημερινή οικονομική κατάσταση. Και να σας πω ότι το Συμβούλιο Εκοφήν θα το γνωρίζετε άλλωστε ασχολείται με τα προβλήματα αυτά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πάνω σε αυτά εξετάζουμε κάθε διαφορετική πτυχή, οτιδήποτε έχει να κάνει και συναντιόμαστε από τον Οκτώβριο πέρυσι στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ, από όταν ξεκίνησε ε, αυτής οι δονήσεις ξέραμε ότι η χρονιά αυτή θα ήταν ακόμα χειρότερη από ό,τι προβλεπόταν και έχουν αλλάξει ριζικά οι μακροπόθεσμες και μεσοπόθεσμες ε, προτεραιότητες και τα όσα κάνουμε. Και τώρα θέλουμε στο ΕΚΟΦΗΝ ε, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σχέδιό της ε, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα προβλήματα που εμφανίζονται στην πραγματική οικονομία γιατί οι οικονομίες ε, είναι ιδιαίτερα αλληλένδετες στις χώρες μας και χάρη και στη νέα κοινή αγορά είναι συγκοινωνούντα δοχεία μπορούμε να πούμε και έχουμε λοιπόν ροή και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη συνεχή γι' αυτό χρειάζονται κοινέ προσπάθειες στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ εξετάζουμε, μελετούμε τους σχετικούς στόχους. Βέβαια πρόωρο είναι ακόμα να δούμε τι, και να πούμε τι θα γίνει με τα μέτρα που εφαρμόζονται στην πραγματική οικονομία αλλά το πρώτο που προσπαθούμε, προσπαθήσαμε και κάναμε έδειξε ότι τα κράτη καταλαβαίνουν βέβαια ε, τον δεινό χαρακτήρα αυτών των προβλημάτων και προσπαθούν να ενισχύσουν ε, την θέση τους. Ε, και εδώ Θέλουμε όλα αυτά ε, να καταλάβουμε ότι εξαρτώνται από ένα άμεσο χαρακτήρα αντίδρασης στην ταχύτητα και χρειάζεται ταυτόχρονα να σεβαστούμε και την αρχή ενός ε, νόμιμου ανταγωνισμού, θεμητού ανταγωνισμού οικονομικού και μιας διαφάνειας όπως το είπε και ο Επίτροπος ε, Αλμούνια στην όλη σημερινή κατάσταση έχουμε μια εκτίμηση για 3% του ΑΕΠ ε, μαζί με τους αυτόματους αυτούς τα θεραπευτές για τους οποίους μιλήσαμε πριν από λίγο και που διαφορετικά, αντρούς, διαφορετικά από ό,τι στις ΗΠΑ παίζουν σημαντικό ρόλο σε εμάς. Αλλά όλα αυτά θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα πριν τα μέτρα όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφραστούν, εμφανιστούν ε, τα αποτελέσματα τα δικά μας οικονομικά. Υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση αδράνεια και θα καθυστερήσει λοιπόν. Θα υπάρξει ακόμα μια περίοδος άσχημων νέων και κάθε μέρα θα έχουμε τα νέα στατιστικά αρνητικά στοιχεία για την όλη πορεία της οικονομίας και βέβαια και για τις διάφορες εταιρείε από πέρυσι. Χρειάζεται όμως να κατανοήσουμε ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε κρίση λαμβάνονται πραγματικά μέτρα. Ξεκίνησαν τα μέτρα από το φθινόπωρο μας πέρασε και βέβαια όλα αυτά για να εκφραστούν οικονομικά μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ε, να μπορέσουμε να αμβλύνουμε κάπως ε, τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης και να εξασφαλίσουμε μια υφόρο ανάπτυξη. Βέβαια δεν θα πρέπει να πιστεύουμε όλοι όλους όσους ε, από τον πολιτικό κόσμο λένε ότι είναι κάτι εξασφαλισμένο αυτό. Η οικονομία της αγοράς ε, προχωράει με κύκλους, κύκλους ανάπτυξης. Ε, δεν υπάρχει κάτι το μόνιμο και σταθερό μια μόνιμη σταθερή πορεία, αλλά εντάξει μπορούμε να εμβλύνουμε τα αρνητικά στοιχεία στους πολίτες μας. Αυτό άλλωστε προσπαθούμε να κάνουμε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και στις χρηματαγορές έχουν ληφθεί επίσης κατάλληλα μέτρα για να μην καταρρεύσει το σύστημα αυτό. Και ε, η λειτουργία μας δεν είναι όπως η συνηθισμένη καθημερινή. Αυτό ισχύει για κάθε τομέα και για τις πιστώσεις που απαιτούνται για μια ανάκαμψη οικονομική και κάθε όθηση οικονομική δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν δεν αποκατασταθεί εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα και έχουμε και ε, είχαμε μιλήσει, είχαμε πει για, τα, για τη βοήθεια στις τράπεζες και επίσης για τα τοξικά οικονομικά προϊόντα. Ε, συζητάμε για αυτά και αυτό κάτι που απαιτείται για ένα θεμητό ανταγωνισμό, σωστό ανταγωνισμό. Αυτά αποτελούν προϋποθέσεις απαραίτητες πραγματικά για, μια, για ένα υγιή ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταλάβουμε και ορισμένες πτυχές σημαντικές που δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να τις αναφέρουμε. Πρώτα απ' όλα, κάποια κράτη δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν παρόμοια παροτριντικά μέτρα όπως μέχρι σήμερα και στο Συμβούλιο Κοφίν οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να το πείσουν και τα δικά τους προβλήματα για να δουν πώς τα κυβερνητικά προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν και τι κόστος απαιτείται για κάτι παρόμοιο που θα μπορούσε κανείς να το αντέξει. Και όλα αυτά δεν είναι εύκολο λογαριασμοί να γίνουν και για διάφορα ε, προϊόντα κίνδυνου κλπ. Εδώ και στο μέλλον θα πρέπει να δούμε πώς θα αποκατασταθεί μια κατάσταση που να διαρκέσει πραγματικά. Εδώ γινόμαστε μάρτυρες ε, μιας μίας οικονομική μας δύναμης, επίσης και μια γύρανση πληθυσμού που θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα στο δημόσιο προϋπολογισμό μαζί με τα συγκυριακά μέτρα τα οποία συζητάμε στο ΕΚΟΦΗΝ για να αντιδράσουμε. Αλλά θα πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη μας και τις μακροπόθεσμες πολιτικές και πώς θα αντέξει μακροπρόθεσμα ο δημόσιος προπολογισμό και πραγματικές βαθιές δραστηριοτικές αλλαγές στο όλο σύστημα λόγω της γύρασης του πληθυσμού. Θα πρέπει να δούμε το συνταξιδοτικό σύστημα και το σύστημα υγείας. και το σύνθημά μας είναι στην Δημοκρατία της Αιχίας Ευρώπη χωρίς εμπόδια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα αυτά τα προστατευτικά που εκδηλώνται καμιά φορά και στα πλαίσια του G7 και του ECOFIN ε, εξετάζονται αυτά. Το ίδιο θα γίνει νομίζω και στο έκτακτο, ε, στην έκτακτη σύνοδο και θα υψώσουμε τη φωνή μας με ένα όχι κατά του προστατευτισμού. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να συναψίσω όσα είπα σε λίγες φράσεις ότι χρειάζεται σε όλες μας τις συζητήσεις να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα μέτρα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά για να αντιδράσουμε από οικονομικής πλευράς. Αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε σε κάθε στιγμή. Και αντιμετωπίζουμε βέβαια και κινδύνους ιδιαίτερες μείωσης του ΑΕΠ μας, επίσης υψηλού ποσοστού ανεργίας, αλλά χρειάζεται να λάβουμε τις ευθύνες των πραξεών μας και είναι δικό μας καθήκον να προχωρήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο ώστε ο κίνδυνος να μην μεταφραστεί σε πραγματικότητα, σε κάτι το πραγματικό. Για να δούμε λοιπόν τι κάνουμε, όπως και για τον προστατευτισμό τον οποίο ανέφερα λίγο πριν. Ο προστατευτισμός είναι αδελφός του παρεμβατισμού και θα πρέπει αντίθετα όλοι μας μαζί να ενώσουμε τη φωνή μας και τα χέρια για να αποφύγουμε παρόμοια μέτρα προστατευτικά να μην αφιερώνται σε εθνικές προσπάθειες τα διάφορα κονδύλια έτσι, πολλές φορές έχουν την τάση να το κάνουν αυτό, να υπόσχονται εθνικά μόνο μέτρα οι πολιτικοί άνδρες, ε, ε πρόκειται για ένα πειρασμό. Αλλά εμείς, ε, έστω και αυτόν είναι εις βάρος του, της, ε, του, του το να είμαστε δημοφιλείς είναι να είμαστε κατά του προστατευτισμού, να μπορούμε να εξηγήσουμε ότι θα ανοίξουμε έτσι το δρόμο με τον προστατευτισμό σε μια πιο βαθιά κρίση από τη σημερινή και ότι ε, χρειαζόμαστε τους γείτονές μας περισσότερο ποτέ και όχι η δική μας μόνο κατανάλωση. Χρειάζεται όλοι μαζί εναρμονισμένα, συντονισμένα να προχωρήσουμε και να απορρίψουμε τον ε, προστατευτισμό. Δεν θα πρέπει να υψώσουμε εμπόδια ανάμεσα στις χώρες μας. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που διατρέχουμε σήμερα. Και ακόμα ένας άλλος κίνδυνος είναι βιαστικών αποφάσεων στις λήψεις μέτρων. Βέβαια με την κρίση καταλάβαμε ότι όσον αφορά εποπτείες και λοιπά των χρηματοαγορών είχαμε κενά εκεί. Αυτό το έδειξε, το απέδειξε η κρίση. Θα πρέπει όμως και είναι μια πρόκληση να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα Χρειάζεται λοιπόν να την περίσουμε την πρόκληση και στην διάσκεψη των 20, των G20 αυτό θα αντιμετωπιστεί και πολλές φορές ε, ε, η δινή κατάσταση όθησε σε βιαστικές αποφάσεις ε, όσον αφορά τη λήψη μέτρων που στο κάτω-κάτω έκαναν περισσότερη ζημιά από ό,τι καλό. Χρειάζεται αυτό το αγκάθι να το αποφύγουμε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε, να πετύχουμε κάτι καλύτερο, μια πραγματική επικοδομητική συζήτηση, να δούμε και τις μελέτες ε, εφικτού τι γίνεται, μια σταδιακή λήψη μέτρων και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αν έχουμε επαναστατικά, βιαστικά μέτρα, τότε σίγουροι σχεδόν είμαστε ότι περισσότερη ζημιά θα κάνουμε από ό,τι όφελος θα έχουμε. Και ακόμα κάτι, ένας ακόμα κίνδυνος που θα ήθελα να τονίσω είναι ο κίνδυνος του τι σημαίνει κόστος για το μέλλον. Δεν διαθέτει ρευστό κανένα κράτος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Έχουμε μόνο τα χρήματα που μπορούμε να δανειστούμε και που θα πρέπει να τα ξεπληρώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και μάλιστα δεν του ζητάμε και την άδεια να το κάνουμε αυτό. Να λοιπόν που αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους της οικονομικής κρίσης και από την άλλη μεριά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο δημιουργούμε να μας κοστίσει πολύ περισσότερο μακροπρόθεσμα λόγω, της, λόγω του χρέους και πώς θα επαναχρηματοδοτήσουμε το χρέος μας και ότι θα μεταβάσουμε το χρέος αυτό στις μελλοντικές γενιές να μην είναι ανυπόφορο το κόστος αυτό για τους όμους των επόμενων γενεών, να μην είναι κάτι που να μπορεί να, να ε, αποφευχθεί. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να μας ε, καταραστούν οι επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, ο Μυροσλάβ Κάλουσεκ, για την δήλωση αυτή. Και τώρα ίσως μπορώ να ζητήσω από τον κύριο Τρισέ να απαντήσει σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων και ερωτημάτων που θα ήθελα να διεξέλθω εντάχει καταρχήν για το θέμα του προστατευτισμού. Εγώ συμφωνώ με την άποψη, την ομόφωνη άποψη που εκφράστηκε εδώ, ότι ο προστατευτισμός σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν πολύ επικίνδυνος. Έχουμε εμπειρίες προστατευτισμού σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας, ήταν τραυματικές εμπειρίες Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε μια οποιαδήποτε μορφή προστατευτισμού στο χρηματοοικονομικό σύστημα, μια αντιμετώπιση μερκαντιλιστική από τα κράτη-μέλη μας και μαζί με την Κομισιόν έχουμε κάνει ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι είναι ισόπεδο το γήπεδο, είναι ίσοι κανόνες ανταγωνισμού, ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Όλες οι προτάσεις λοιπόν για την ανάκαμψη του συστήματος θα το λάβουν αυτό υπόψη. Επίσης θεωρούμε ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι ουσιώδες να διατηρηθεί. Οι κανόνες του έχουν τροποποιηθεί πριν από μερικά χρόνια ακριβώς για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε σήμερα ενώπιόν μας. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό να παρακάμψουμε το σύμφωνο σταθερότητας και να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι κανόνες του συμφώνου λένε ότι όταν υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καταρχήν την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Και αυτό βασίζεται στην αντίληψη ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι οικονομικές συνθήκες είναι βιώσιμες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να χαράξουμε τις κατάλληλες πολιτικές για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τα συμφέροντα των επερχομένων γενναίων. Για το τρίτο σημείο τώρα το οποίο αναφέρθηκε που είναι μια αντικυκλική πολιτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε εγώ θέλω να επιβεβαιώσω ότι θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο της κάθε μεγάλης μονάδας σε παγκόσμιο επίπεδο να αναλάβουμε αντικυκλική δράση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μπούμε σε δεύτερη φορά σε μια κατάσταση όπου εμείς ενισχύουμε τους κύκλους οικονομικούς την ταχεία ανάπτυξη και την ταχεία κατάρρευση λοιπόν που μπορεί να προκύψει από την ενίσχυση των κύκλων, εγώ τονίζω πάντα ότι η ανάπτυξη πρέπει να ξεκινάει στο σπίτι μας, στην κάθε χώρα μας. Ο ανταγωνισμός μέσα στην Ευρώπη αλλά και μέσα σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποφασιστικό. Να αυξάνει την παραγωγικότητα κατά μοναδιαίο μοναδία μονάδα εργασία. Πρέπει όλοι μας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε προσεκτικά τις πολιτικές ανταγωνισμού οι οποίες ακολουθούνται στα κράτη μας. Θα απαντήσω επίσης και στην απάντηση η οποία διατυπώθηκε για το γεγονός, όπως είπε ο κύριος Γκέμπελς, οι τράπεζες δεν μεταβιβάζουν πάντα τη μείωση των επιτοκίων που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στους καταναλωτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά και να υπάρχει απαραίτητη υποπτία. Βέβαια, δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να λέμε στις τράπεζες ότι φταίξατε γιατί πήρατε πάρα πολλούς κινδύνους και μετά τους λέμε φταίτε γιατί φοβόστε σήμερα να αναλάβετε κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια λογική αντιμετώπιση και κλείνοντας θα έλεγα ότι το μήνυμα το οποίο θέλω σας μεταφέρω είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την βραχυπρόθεσμη κατάσταση και τις προκλήσεις που έχουμε τώρα, που είναι κάτι το πολύ επιτακτικό και καταπήγον, αλλά συγχρόνως διατηρώντας μια εικόνα στον ορίζοντα του μακροπρόθεσμου. Και αυτό έρχεται από την κοινή λογική. Πρέπει να φροντίσουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας ακόμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην επίλυση των προβλημάτων μας, γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας στην επίλυση προβλημάτων που αποτελεί το θεμελιώδες στήριγμα της εμπιστοσύνης σήμερα. Η σημερινή εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών είναι το πιο σημαντικό αλλά και το πιο σπάνιο αγαθό που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την αηφορία, να έχουμε πολιτικές οι οποίες έχουν αηφόρο χαρακτήρα, να μην ξαναγυρίσουμε στο status quo άντε και ούτε να δράσουμε σε επίπεδο μεμονωμένο και αποσπασματικό σαν μεμονωμένα κράτη. Αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε την μακροχρόνια σταθερότητα για να επιλύσουμε τα σημερινά προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τρισέ. Και τώρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Hans Kert Πέτερινγκ. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σεράου για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και θα ήθελα να πω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περατώσει τη διαδικασία κύρωσης. Παραμένει μοναχα η υπογραφή του Πρόεδρου της Πολωνίας και τα δύο νομοθετικά σώματα στην Πολωνία έχουν εγκρίνει τη συνθήκη και είναι εύλογο ότι θα πρέπει να υπογραφεί και από τον Πρόεδρο της Πολωνίας η συνθήκη. Πρέπει να υπογράψει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας γιατί εκκρεμεί ακόμα μια διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα μπορεί να υπογράψει τη συνθήκη ο πρόεδρο τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Επομένως και στην Πολωνία και στη Γερμανία νομίζω πηγαίνουν καλά τα πράγματα και έχουμε ακόμα και την ψηφοφορία πρέπει να γίνει στην άνω και κάτω ε, Τσεχική Βουλή. Οι Τσέχοι συνομιλητέ μα ίσω θα να προσθέσουν κάτι για το θέμα αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να του παροτρύνω να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε κάτω από τσεχική προεδρία να μπορέσει στην Τσεχία να εγκριθεί η συνθήκη της και τέλος έχουμε το δημοψήφισμα το οποίο εκρεμεί στην Ιρλανδία. Ελπίζουμε ότι η Ιρλανδία θα δώσει και αυτή στο επερχόμενο δημοψήφισμα την συγκατάθεσή της. Επομένως, εν κατακλείδη, μία αποτυχία της συνθήκης της Λισαβόνας θα είναι σε πολιτικό και ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο μια αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας αυτή την αποδυνάμωση, αντίθετα θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι εάν υπονομευθεί η συνδίκη της Λισαβόνας, αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει κανείς και την ευθύνη να μην υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να είμαστε προς μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου, αλλά μια ισχυρή δημοκρατική και διάφανη ένωση. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι πρέπει να μπει σε εφαρμογή των αδεχείων των δυνατών συνδίκης Λισαβόνας. Ευχαριστώ ο κύριος Ράινχαρτ από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον Πρόεδρο για τη διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης με κεντρικό θέμα το New Deal στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν πολύ, μια πολύ εύστοχη επιλογή αυτού του θέματος και σας συγχαίρω και πάλι. Όπως ελέγχθη, ο κόσμος μας έχει γίνει ένα παγκόσμιο χωριό και οι προκλήσεις σε οικονομικό επίπεδο είναι ήδη πανευρωπαϊκοί τα θέματα των ε, ratings της ε, βαθμολόγησης της ε, δανειοληπτικής ικανότητος, το να υπάρχουν κοινά στάνταρ στη λογιστική είναι κοινά προβλήματα και σίγουρα είναι πολύ σημαντική η αντιμετώπιση του να μην δεχτούμε τον προστατευτισμό από τη δική μου χώρα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε ένα κοινό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζωγόνηση της οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να μπορέσουν να προχωρήσουν πολύ σημαντικά. Περιμένουμε στο πρώτο τέταρτο του 2009 μια κάμψη κατά 3 ως 4% της οικονομικής δραστηριότητας. Εγώ δεν θεωρώ ως λυσιτελές ότι προγράμματα που αφορούν παραγωγός χάρη την ενέργεια ή τις ευρυζωνικές συνδέσεις στις τηλεπικοινωνίες να προχωρήσουν χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση και να μην μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα προγράμματα υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τα χρήματα θα πάνε σε άλλες επενδύσεις. Θα πρέπει να τονίσω την αρχή της λιτότητας και της πειθαργίας του προϋπολογισμού και επομένως τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δαπανηθούν σε στόχους οι οποίοι δεν είναι χρήσιμοι για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα σε στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν αμέσως και το ταχύτερο δυνατό. Έχουμε μειώσει επίσης και τις διαδικασίες, έχουμε διαδικασίες μάλλον τις ε, προθεσμίες για τις ε, προμήθειες σε 30 μέρες από 60 ε, μέρες και παραπάνω. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να επιταχύνουμε πάρα πολύ τις διαδικασίες για, την, για τους διαγωνισμούς, για τα προγράμματα ανάκαμψης και έχουμε επίσης αυξήσει και τα όρια για αυτούς τους ταχύς διαγωνισμούς σε 10 εκατομμύρια, αυτό θα ευνοήσει την ταχεία ε, ανάληψη έργων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και επομένω θα βοηθήσει την ανάκαμψη. Επίση, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε και κατάλληλη στοχοδεσία για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πρέπει να έχουμε ένα στόχο 25% μείωση, να αναφέρει σε τι ο Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραβιαστούν οι κανόνες διαδικασίες. Είναι χρήσιμο να υπάρχει ένας φορέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορεί να παρακολουθήσει το κόστος της γραφειοκρατίας, να βρει τους τρόπους με τους οποίους θα μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει καλύτερη νομοθεσία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει η δυνατότητα να βαπτίζονται ως ευρωπαϊκά πρότυπα μία σειρά από διαδικασίες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει με μία τέτοια κατεύθυνση στη Βάδη Βιρτεμβέρη και αυτό θα μπορούσε να μεταλαμβαδευτεί και σε άλλες περιφέρειες Ευρώπης αλλά και πάλι θέλω να σας συγχαρώ γιατί μας δίνεται αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το πιο σημαντικό θέμα της σήμερα ημέρας. Σας ευχαριστώ. κυρία Πέτερσον από το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας. Της Λετωνίας, συγγνώμη. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Τσεχικό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας δίνουν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η Λετωνία ελπίζει ότι η κρίση δεν θα οδηγήσει τελικά στην ε, απώλεια της βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό ευχαριστώ όλα τα κράτη-μέλη για την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν δηλαδή, μέσω της στήριξης της πρότασης της Κομισιόν για χρηματική βοήθεια και προς τη Λετωνία η οποία αντιμετωπίζει βαθιά κρίση. Και τώρα ένα σχόλιο για το τι αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς ίσως αυτό να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους που θα αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση. Η ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση είναι πολύ σημαντική για την ανάκαμψη της οικονομίας μας διότι τον Δεκέμβριο η Βουλή μας δέχτηκε έναν πολύ αυστηρό προϋπολογισμό για το 2009. Στη χώρα μου η ανάπτυξη μειώθηκε από 10 σε 5% και γι' αυτό είχαμε την επιλογή είτε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας, το ΛΕΤ, είτε να κάνουμε άλλες, άλλου είδους δαπάνες, νέες δαπάνες. Αυτό επιλέξαμε τελικά. Από 18% τις αυξήσαμε σε 20% και αυτό δημιούργησε πολλές αντιδράσεις αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε ταυτόχρονα να εφαρμόσει ένα σχέδιο ανάκαμψης και ένα σχέδιο διασφάλισης μακροοικονομικής σταθερότητας. Αυτό δεν ήταν εύκολο διότι έχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει και για την έρευνα και για την αγορά της εργασίας και για το εμπόριο και για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτά τα δύσκολα καθήκοντα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε παρά αν υπάρξει και μια θεσμική αναδιοργάνωση και μειωθεί και το γραφειοκρατικό άχθος και όλα αυτά σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όταν ψάχνουμε λύσεις σε κρίση δεν πρέπει να ξεχνάμε τα υπάρχοντα εργαλεία. Ελπίζουμε ότι όταν τα οικονομικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ότι δεν θα ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να σταματήσει η αρνητική μας μέχρι τώρα πορεία. Έχουμε επίσης αυξήσει τα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία και γενικότερα σχεδιάσαμε 2,4% του ΑΕΠ να διαθέσουμε για την αναθέρμανση της οικονομίας. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματα στη Λετωνία. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου και επίσης άμεση και γρήγορη αντίδραση από το Κοινοβούλιο και ικανότητα λήψης μη δημοφιλών αποφάσεων. Σήμερα στην Ένωση καταλαβαίνουμε ως Λετωνή πολιτική ποιες είναι οι ευθύνε μας αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα έχουν πολιτικό κόστος. Είναι όμως παρήγορο να βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνοι μας την κατάσταση και σας ευχαριστούμε για όσα έχετε κάνει για τη Λετωνία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάτεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος μας αναφέρθηκε ήδη στη συνθήκη της Λισαβόνας και θα ήθελα να τονίσω την σημασία αυτής της συνθήκης και η Λισαβόνα παίζει στην καθημερινή ζωή ένα σπουδαίο ρόλο. Αποφάσισαν ε, ότι σε 10 χρόνια η ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι η πιο δυναμική που θα βασίζεται στη γνώση. Εδώ και 9 χρόνια έγινε αυτό. Κανονικά σε ένα χρόνο θα έπρεπε όλα αυτά να τα έχουμε πετύχει. Είχαμε πει τότε οι ηγέτες κρατών κυβερνήσεων σε 10 χρόνια ότι θα γινόταν. Και με τις οδηγίε της Λισαβόνας τότε ο καθένας χαιρόταν για τις αποφάσεις αυτός των ε, ηγετών κρατών και κυβερνήσεων για μια νέα δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η διαπίστωση ήταν ότι εν μεταξύ δεν έγινε τίποτα για να εφαρμοστούν αυτά στην πραγματικότητα και να εμφανιστούν στην πραγματικότητα. Εντάξει, για τη στρατηγική τη Αβώνας αυτή αναφέρθηκε, τονίστηκε κλπ. Αλλά τίποτα κενή, χωρίς πραγματικό περιεχόμενο και ουσιαστικά η Λισαβόνα ε, εκπροσωπεί πια, συμβολίζει λόγια, λόγια, λόγια, αλλά όχι πράξεις, όχι ενέργειες. Και εδώ λοιπόν όλα, ε, όλα αυτά για την εφαρμογή προκαλούν δημιουργούν προβλήματα. Βλέπουμε και την έκφραση ενός κάποιου προστατευτισμού. Το ακούσαμε και σήμερα αρκετές φορές ε, και για την παρεμβοτισμό των κρατικών στην οικονομία. Εντάξει, θέλει κανείς να ανοίξει ένα δρόμο, αλλά μήπως πρόκειται για μια οπισθοδρόμηση εδώ ε, απέναντι στην κρίση από πλευράς δημοσίου κλπ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που γεννιέται και το μέλλον επίσης θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από όλα αυτά. Εντάξει, η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν καλή. Επέτρεπε στην ευρωπαϊκή οικονομία να ευθυγραμμιστεί με την αμερικανική και με τις ασιατικές οικονομίες. Αν θέλουμε πραγματικά ε, νέες θέσεις απασχόληση, μια υφόρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε μια νέα δυναμική που θα βασίζεται στη γνώση. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε απέναντι στην κρίση αυτή, να προσέξουμε αυτή την οικονομία ε, πώς θα την τονώσουμε μέσω καινοτομιών. Μια οικονομία που να αποκρούει όλα τα χτυπήματα να τα αντέχει. Χρειάζεται μια στρατηγική έξυπνη για να ενισχύσουμε την οικονομία μας και απέναντι στους υπόλοιπους. Είναι η σημερινή ευκαιρία και το είπε ο Σνάριφος Γκέμπελς και μάλιστα πολύ σωστά. Είναι οι χώρες αυτές που ε, συνέλαβαν την ιδέα της στρατηγικής της είναι και τα κράτη που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτής της Αβώνας. Είναι και σωστή αυτή η παρατήρηση. Στο μέλλον τι θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να περάσουμε μήπως σε μια οικονομία που θα χαρακτηρίζεται από μια ισχνή κατανάλωση, χαμηλή κατανάλωση και χωρίς ε, ε χρήση ε, άνθρακα πανασχάρη και να δούμε τις κλιματικές αλλαγές, όλα αυτά χρειάζεται να δούμε τη στατική της αβώνας. Οι διάφορες αναλύσεις που έγιναν ήταν και σωστές οι κατάλληλες, είναι πάντα επίκαιρες, ανταξύ όμως δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα, πρέπει όμως να καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Επιτέλους θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εκφράσουν και κατάλληλα την καλή τους θέληση και μας έδωσε και το παράδειγμα, θα πρέπει να μας δώσει το παράδειγμα και η Επιτροπή. Έχουν, ε, έχει ε, επιδειχτεί κάποια θετική αντιμετώπιση. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε τώρα εδώ παθητικοί και να μην κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει κάτι να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αϊβαλιώτης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της συζήτησης και να συγχαρώ και όλους τους ε, συμμετέχοντες για το ότι αναφέρθηκαν πολύ συχνά, το άκουσα, στην γύρανση και στην υπογεννητικότητα. Και επίσης συγχαρητήρια χρειάζονται, αξίζουν σε αυτούς που συνέταξαν το General Documentation αυτής της ε, συζήτησης που πάλι αναφέρεται στη γύρανση και στην υπογεννητικότητα. Τα λέω αυτά επειδή όποιος διάβασε το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2009 θα είδε ότι ούτε μία φορά δεν υπάρχει αναφορά στη γύρανση και στην υπογεννητικότητα. Και πρέπει να σας πω ότι ως Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων λάβαμε ομόφωνη απόφαση να διαμαρτυρηθούμε στην Κομισιόν για την παντελή έλλειψη αναφοράς στην υπογεννητικότητα και στη γύρανση στην Ευρώπη όταν είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης σβήνει. Μιλάμε για ένα New Deal και θα ήθελα έτσι να επικεντρωθώ στα κριτήρια του Maastricht, στο Σύμφωνο Σταθερότητας, γιατί είναι ασφιχτικά και, για πο πολλές χώρες τραγκαλίζονται από αυτά τα κριτήρια. Ο κύριος Λένε αν θυμάμαι καλά, ανέφερε ότι υπάρχει ευκαμψία ή θα πρέπει να υπάρχει ευκαμψία στο Σύμφωνο Σταθερότητα. Πρέπει να τη δούμε αυτή την ευκαμψία. Προέρχομαι από μια χώρα η οποία έχει τι μεγαλύτερε κατακεφαλήν αμυντικέ δαπάνες στην Ευρώπη. Το 5% του GNP, του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της Ελλάδας, πηγαίνει σε αμυντικέ δαπάνες, διότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει το βάρος της τουρκικής επιθετικότητας, του τουρκικού εθνικισμού. Έτσι λοιπόν είναι μια χώρα η οποία έχει τεράστιες αμυντικέ δαπάνε, δεν είναι η μόνη, η Ελλάδα όμω είναι η χώρα με τι βαρύτερε αμυντικέ δαπάνε κατά κεφαλή και παράλληλα έχει να τη ρίση και τι προβλέψει, τι ασφιχτικέ, επαναλαμβάνω προβλέψει του Συμφώνου σταθερότητα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα κριτήρια, πρέπει να χαλαρώσουν. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να θέσω είναι τα τεράστια ποσά που προβλέπει ο κοινοτικό προπολογισμό για χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εδώ μπροστά μου ένα επίσημο έγγραφο τη Κομισιόν με τον αριθμό 3917 του 08 αυτό το έγγραφο αναφέρει τα ποσά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι άνθρωποι που μας ψηφίζουν, οι φορολογούμενοι που μας στείλανε στις Εθνικές Βουλές και εσάς τους Ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί φορολογούνται και βλέπουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από το 1992 ως σήμερα στην Τουρκία και στα Σκόπια. Σε χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα αντιμετωπίζουμε μια κρίση Είπε σωστά πριν ο κύριος Παπουτσής ότι πρέπει να υπάρξει επένδυση Στη, στη, πρέπει να επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να υπάρξει επένδυση σε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, να μειωθεί η ανεργία. Πολύ σωστά το ανέφερε αυτό. Μήπως πρέπει να μείνουν εδώ αυτά, ε, όταν λέω εδώ εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υπάρξει και η αντίστοιχη θετική ε, αντίδραση από αυτές τις χώρες προς τα, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουν και οι φορολογούμενοι τους επιβαρύνονται για να παίρνουν αυτοί 13 δισεκατομμύρια ευρώ επαναλαμβάνω στην Τουρκία και στα Σκόπια. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σπαντώνη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο και την Τσεχική Προεδρία που οργάνωσαν αυτή την πολύ σημαντική διακοινοβουλευτική συνάντηση. Συνάδελφος εκπρόσωπος της Ιταλικής Γερουσίας, συμφωνώ με εσά το ότι απαιτείται προσπάθεια να ανακουφιστεί ο πληθυσμός σε μια σοβαρή κρίση και στην Ιταλία και αλλού λόγω των ειδικών διορθωτικών χαρακτηριστικών που έχει. Αλλά προϋπόθεση και είδαμε και στις Βρυξέλλες να υπάρχουν ανησυχίε για πειρασμό προστατευτισμού θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να τονίσω ότι σημερινή οικονομική κατάσταση φαίνονται να είναι ανεπαρκείς οι κανόνες για την οικονομία και τις χρηματαγορές. Ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός χρειάζεται ένα νέο Bretton Woods για ένα νέο αρχιτεκτόνημα του καπιταλισμού της τρίτης γενιάς. Αν θέλουμε αυτή η κρίση να μην οδηγήσει σε εσωτερική έκρηξη του εύθραυστου διεθνούς συστήματος νέες συμφωνίες να είναι δημοκρατικές, να μην είναι μόνο μια συμφωνία μεταξύ μεγάλων, να ληφθούν υπόψη και η κοινωνία των πολιτών, τα διάφορα δίκτυα, οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι. Θα ήταν λάθος να έχουμε μια διαχείριση της αγοράς και της συγκυρίας που θα προσπαθήσει να λύσει μια παγκόσμια κρίση καλώντας μόνο τους διεθνούς ηγέτες για να γράψουν νέους κανόνες. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να μην μου αρέσει το ότι δεν έγινε αποδεκτή μια πρόταση της τελικής κυβέρνησης να εγκριθούν να υιοθετηθούν προγράμματα κατά της κρίσης που να διαχειρίζονται άμεσα τα όργανα της Ένωσης και αντίστοιχε υποδομές. Εγώ είμαι φιλοευρωπαίστρια. Μου είπαν ότι αυτό δεν γίνεται για λόγους οικονομικούς. Ερωτώ, είναι δυνατόν να μην μπορεί να βρεθεί μια λύση με την υποστήριξη όλων των κρατών μελών για μια πολιτική πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή, για μια μακροπολιτική. Γιατί να μην στηριχτούμε σε προγράμματα και κινητοποίηση πόρων χωρίς να χρησιμοποιούμε τη δύναμη της Ένωσης και το δυναμικό του ευρώ ως αποθυματικού νομίσματος. Η Ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε μια σειρά μέτρων σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης. Δεν θα σας κουράσω απαριθμώντας τα μέτρα αυτά, γιατί ξέρω ότι χρόνο δεν έχουμε. Θέλω μόνο τελειώντας να πω το εξή. Η Ευρώπη από την κρίση θα βγει μόνο αν οι σημερινέ χρηματοπιστωτικές θύελες, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτική, δεν είναι κρίση της αγοράς εργασίας, είναι και του κοινωνικού κράτους. Πολλαπλή κρίση. Με ένα νέο σύμφωνο, μια νέα συμμαχία μεταξύ της κοινωνίας, των κυβερνήσεων, των προσώπων που να εξασφαλίζει ένα επαρκές εισόδημα για την καθημερινή δουλειά των ανθρώπων. Εύχομαι οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να συνδυάσουν ευελιξία και σοβαρότητα με σεβασμό των μελλοντικών γενιών. Σας ευχαριστώ όλους σας που με ακούσατε. Πρόεδρος, η κυρία Χάρμς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, όταν μιλάμε για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και πολιτισών στην διαχείριση της κρίσης, καταρχήν δεν πρέπει να νομίζουμε ότι αυτή η κρίση έχει δημιουργηθεί από τα έξω εμείς έχουμε εμπλακεί ως Ευρωπαίοι στην δημιουργία αυτής της κρίσης, η οποία είναι τμήμα της στρατηγικής της αγώνας. τμήμα της στρατηγικής απορρίθμισης των τελευταίων δεκαετών και που έχει συντείνει στην κατάρρευση των χρηματοοικονομικών αγορών. Θα πρέπει τώρα να περιμένουμε μια πιο αυτοκριτική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήδη είχε συν... σήματα της κρίσης από το 2007, θα μπορούσε ήδη να είχε αντιδράσει και παρά το γεγονός ότι έγιναν πιο έντονα αυτά τα μηνύματα κινδύνου δεν υπήρξε καμιά αντίδραση, δεν υπήρξε καμιά κίνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών. Και επίση είναι λαθασμένο, νομίζω και πολύ κοντόφθαλμο να νομίζουμε ότι είναι μια κρίση μονάχα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Όπω είπαμε πολλοί συνάδελφοι, έχουμε τρει κρίσει συγχρόνω. Έχουμε και την κρίση σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί έχουμε μια βαθιά ρήξη και ένα βαθύ διχασμό, διχασμό στις κοινωνίες μας, μια ανισοκατανομή του εισοδήματος. Έχουμε λοιπόν και την κρίση αυτή σε επίπεδο κατανομής εισοδήματος και έχουμε επίσης και τα προβλήματα της κρίσης του περιβάλλον που οφείλονται σε μια λανθασμένη οικονομική κατεύθυνση που έχει οδηγήσει σε υπερκατανάλωση. Έχουμε λοιπόν προσπάθειες να παρέμβουμε με εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ε, ευρώ, αλλά αυτό σημαίνει πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις τρεις κρίσεις παράλληλα. Δεν χρειαζόμαστε ένα New Deal, χρειαζόμαστε ένα πράσινο New Deal, το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις τρεις κρίσεις συγχρόνως, με μία συνεκτική αντιμετώπιση. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μία εθνική εγωιστική αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Θα ήταν πολύ καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν ισχυρότερη και να μπορούσε να δράσει συνολικά και να δράσουν όλοι από κοινού. Χρειαζόμαστε εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να επιτύχουν να συμφυλατήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου τα επισκιάζει όλα η συζήτηση για την ε, Λισαβόνα και τις συνθήκες της Λισαβόνας. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις αμφιβολίες για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το να δούμε ήδη τι έχουμε κάνει με τη στρατηγική της Λισαβόνας στο παρελθόν. Εάν έχει ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση, αν πραγματικά ήταν σωστή αυτή η αντιμετώπιση της ε, ε, διαδικασίες της Λισαβόνας και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα έχουν έρθει από έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν σκεφτούμε λοιπόν τι έχει γίνει μέχρι τώρα θα έχουμε ίσως μια πιο κριτική στάση απέναντι στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λάρσεν από το Δανίκο Κοινοβούλιο θα λάβει το λόγο. Ναι. Αντιμετωπίζουμε μία δινή κρίση στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, βέβαια δεν χρειάζεται να μας καταλαμβάνει πανικός. Ε, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύουμε πνεύμα δραστήριο με διάθεση λήψης αποφάσεων να προχωρήσουμε δηλαδή σε συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν θα πρέπει η ευρωπαϊκή σταθερότητα να τεθεί σε κίνδυνο. Χρειάζονται λύσεις Χρειάζονται λύσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα νέα προβλήματα και δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε καινούργια προβλήματα και βράχει πρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα ταυτόχρονα. Χρειάζεται να διατηρηθούν λειτουργούντες ε, μηχανισμοί και σε κοινωνικό επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την οικονομία αγορά στην κοινωνική και θα πρέπει να αποφύγουμε οποιονδήποτε πανικό. Οι μηχανισμοί αυτοί έδειξαν ότι μέχρι τώρα υπήρχαν σταθεροποιητές καλοί στην ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει να διατηρήσουμε σταθερή την πορεία μας προς τα εκεί για αυτή την επίλυση των προβλημάτων. Θα πρέπει να αποφύγουμε ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή προστατευτισμού. Δεν γίνεται να δεχτούμε τον προστατευτισμό γιατί θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα ιδιαίτερα άσχημα, ιδιαίτερα σοβαρά και θα μας οδηγούσε σε μια εποχή πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί να δει να επαναλαμβάνεται. Είναι σημαντικότατο λοιπόν, ε, έχοντας συνείδηση το τι συμβαίνει, να ενεργήσουμε και θα πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε την καταλληλότερη στιγμή με τα καταλληλότερα μέσα. Γι' αυτό ακριβώ σημαντικό είναι πάντα να δούμε τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον κόσμο τώρα τελευταία. Το 2050 ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θα είναι μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού και αυτή η πρόκληση είναι τρομερή. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε πρωτοβουλίες για τη σταθερότητα και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα. Θα πρέπει να διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα εδώ στην Ευρώπη. Χρειάζεται μία ανανέωση. Τι εννοώ. Οι προσπάθειες τις οποίες καταβάλουμε στην Ήπειρό μας ε, και στην Ευρώπη ακριβώ θα πρέπει να επικεντρωθούν πάνω στην ενέργεια, στην ενέργεια την πράσινη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι κάτι το πολύ σημαντικό λόγω της καταστάσεως που επικρατεί στον, ε, για το κλίμα, στον κόσμο ολόκληρο και στην Ευρώπη και επίσης ε, να έχουμε διαθέτουμε μια οικονομία που να βασίζεται στην γνώση. Εδώ και αρκετά χρόνια στη Δανία σημειώνουμε πρόοδο χάρη στην Flexi Security η οποία ισχύει στην αγορά εργασία στη Δανία και ελπίζουμε να μην μας παρεμποδίσει η υπόλοιπη Ευρώπη και να μην είμαστε οι μόνοι που θα το υιοθετούμε αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Ράχελ από την, το Κοινοβούλιο της Αυστρίας. Έχετε το λόγο. Ich glaube, es wurde heute schon viel Richtiges gesagt. Θα ήταν καλύτερο να είχαμε πει σήμερα να σκεφτούμε ποια είναι τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε τώρα και είναι απαραίτητα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρώτα απ' όλα η Ευρώπη είναι μια παγκόσμια δύναμη. Δεν έχει μονάχα ευθύνη για τον εαυτό της, έχει ευθύνη και για, άλλες, για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και τις χώρες στα έξω σύνορά μας, στη γειτονιά μας, που χρειάζονται και αυτές κάποια βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή και να αποφύγουν την ε, ένδια. Υπάρχουν χώρες όπως η Ουκρανία, η Κροατία, οι οποίες χρειάζεται να βοηθηθούν για να μπορέσουμε και εμείς μετά από την κρίση να ευνοηθούμε από τη δική τους παρουσία στα ε, όρια της Ευρώπης. Επίσης θεωρώ ότι θα είναι μεγάλος κίνδυνος να υπάρξει παραβίαση του Συμφώνου σταθερότητα με υπερβολικά ελλείμματα στι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό περιμένω από την Κομισιόν το ταχύτερο δυνατό και με αυστηρό τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ελλείμματα για να υποστηρίξουν τι βιομηχανίε του που βρίσκονται σε κρίση. Αλλά αυτά θα οδηγήσουν σε ένα φαινόμενο ντόμινο. Θα οδηγήσουν σε μια ανάλογη κατάσταση και τι άλλε χώρε και επομένω, το αποτέλεσμα θα είναι να αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη με εκτύπωση χρήματο τα υπερβολικά χρέη τα οποία θα, δημιουργήσει, θα έχουν δημιουργήσει. Τρίτον, θα πρέπει να έχουμε και κάποιο οραματιστικό χαρακτήρα. Για μένα είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κοινωνία γνώσης η οποία λειτουργεί ακόμα με βάση μια κοινωνία η οποία έχει ακόμα ένα κυρίως βιομηχανικό χαρακτήρα. Εμείς θέλουμε να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι θα είναι με υψηλά προσόντα και με υψηλές γνώσεις. Και επομένως θα πρέπει αντί να ευνοούμε μονάχα αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στο χρηματοοικονομικό τομέα και να τους δίνουμε υψηλά πριν, θα πρέπει να βοηθήσουμε να ανέλθουν στην εξουσία και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινωνικές δεξιότητες και μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Επίσης, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η μείωση της γραφειοκρατίας που είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνει ως ρεφρέν πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελαφρύνει το άκρο των επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν 10 εργαζόμενους, 3 τρεις εργαζόμενους και πρέπει να καταδαπανούν το 10-20% του χρόνου τους για να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις τις επιβαρύνει τα μάλα. Θα πρέπει και αυτό το στοιχείο λοιπόν η Κομισιόν να το λάβει υπόψη της για την αντιμετώπιση γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσίμερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και εγώ κύριε Πρόεδρε θα μπορούσα να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε η κυρία Χάρμς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί νομίζω ότι τίθεται το ερώτημα τι ρόλο έχει παίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την όξυνση της κρίσης. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε από κατά μέρο και να θεωρήσουμε ότι όλα έχουν προκληθεί από εξωτερικού παράγοντε. Και εμεί έχουμε συμβάλει ω Ευρωπαϊκή Ένωση στη δημιουργία αυτή τη κρίση και αντίθετα με άλλου συναδέλφου, εγώ νομίζω ότι και η στρατηγική τη Λισαβόνα έχει διαδραματίσει ένα ρόλο στην όξυνση τη κρίση. Δεν έχει εμποδίσει την κρίση όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι. Γιατί το δόγμα της απεριόριστης ελευθερία κίνηση του κεφαλαίου που έχει υποστηριχθεί με την παροκρουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει καθαγιαστεί στην συνθήκη της Νίκαιας και προσεχώς και στη συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης ενώ βλέπουμε σήμερα ότι τα διεθνή χρηματοοικονομικά όργανα θέλουν να περιστύλουν αυτή την αλόγιστη ελευθερία. Επίσης, τα προγράμματα ανάκαμψης στα συγκυριακά στα κατημέλια από μία άποψη είναι θετικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, εφόσον εξυπηρετούν τη στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει στο παρελθόν, δεν πρόκειται να επιλύσουν το πρόβλημα. Θα ήθελα επίση να ζητήσω από την Κομισιόν να τροποποιήσει τη θέση της, γιατί η αντιμετώπιση της μέχρι στιγμής είναι κατευθυνόμενη μονάχα στι χρηματα... στις χρηματαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί και η εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όχι μόνο να αντιμετωπίσει τα θέματα σταθερότητα των τιμών, αλλά να εξασφαλίσει και την σταθερότητα των συστημάτων ε, πληρωμών, τα συστήματα ε, ε, να υπάρχει σεβασμός των ρυθμίσεων και οι τράπεζες να σέβονται τους εθνικούς και τους διεθνείς κανόνες και να υπάρχει δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που υπάρχει πάυση πληρωμών από τράπεζες. Επίσης, Νομίζω ότι οι δράσεις διάσωσης και τα εθνικά προγράμματα ε, ανάκαμψης θα πρέπει να μην περιοριστούν σε μεμονωμένες ενέργειες, θα πρέπει όλα αυτά να στοχεύουν σε μεγαλύτερες επενδύσεις του δημόσιου τομέα και δημιουργία δομών στο μέλλον, ώστε να απεφευχθούν στο μέλλον τέτοιες κρίσεις και να εμποδίσει την σειρά παραγόντων την διασύνδεση των παραγόντων που έχουν οδηγήσει σε μια κρίση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μην γίνει αυτό με περαιτέρω ε, επιβάρυνση της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ο χρόνος για τη συζήτηση έχει λήξει, ο χρόνος που είχαμε, όσοι δεν πήρατε μέρος στη συζήτηση σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε κατά προτεραιότητα αύριο. Τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο Πέτερινγκ. Χρήσιμο είναι να ξέρετε ότι αύριο θα συνεχίσουμε. Αυτοί οι οποίοι είναι στον κατάλογο λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν το λόγο. Σας λέω μονάχα μερικά πρακτικά και διαδικαστικά θέματα. Η ομάδα εργασία 1. Πρόθεση των επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, το επιχειρήν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσει την εργασία της εδώ σε αυτή την αίθουσα. Η ομάδα εργασίας 2 Κοινωνική Ευρώπη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης Αντιμετώπισης Ένδυας Ελευθερία Διακίνησης απέναντι στην αίθουσα 3 σε 50. Απλώς βγαίνετε και πηγαίνετε στην απέναντι αίθουσα. Και η τρίτη ομάδα εργασίας για την αηφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη, αηφόρο ανάπτυξη και προστασία του, του κλίματος. Στον όροφο 1 κατεβαίνετε δύο πατώματα λοιπόν με τις σκάλες και είναι η αίθουσα 1α002. Κάτι ακόμα πιο ευχάριστο, αλλά και η εργασία μας είναι τρομερά ευχάριστη. Στις 19 και 10 θα λάβει χώρα ένα κοκτέιλ στο άλλο κτίριο, στο κτίριο ΑΣΠΕ, Αλτιαροσπινέλη δηλαδή, το οποίο είναι απέναντί μας από την Πασαρέλα. Θα δείτε ένα μεγάλο άγαλμα το οποίο μας έρχεται από την προηγούμενη Ιταλική Προεδρία. Θα έχουμε λοιπόν ένα κοκτέιλ στις 19 και 10 στο εστιατόριο των ε, βουλευτών στις 19 και 45 και εκεί σας καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βραδινό δείπνο σας εύχομαι καλές διαβουλεύσεις και θα βρεθούμε στο κοκτέιλ και στο δείπνο και αύριο ξεκινούμε το πρωί στις 9 και 30. Ευχαριστώ πολύ.